Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί παρευρισκόμενοι και όσοι μας παρακολουθείτε παντού στην Ευρώπη. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, Ελένα Ντάλη, σας καλωσορίζω θερμά. Είστε η υποψήφια επίτροπος για την ισότητα και έχουμε εδώ την κοινή ακρόαση που συμπροεδρεύω με την κυρία Ντούρις Νικολσόνοβα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που συνδέεται με αυτή την ακρόαση εκπροσωπείται εδώ. Είναι μεγάλη επιτυχία που θα έχουμε μία επίτροπο ειδικά για θέματα ισότητας στο μέλλον. Είναι κάτι καινούριο στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Πριν αρχίσουμε την ακρόασή μας, υπενθυμίζω ότι με βάση τις καθεντήρες γραμμές για την έγκριση των επιτρόπων, το παράρτημα 7 του εσωτερικού κανονισμού, το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους υποψηφίους επιτρόπους στη βάση των ε, γενικών προτεραιμάτων τους, της ε, δέσμευσής τους για την, ε, το ευρωπαϊκό εγχείρημα και την προσωπική τους ανεξαρτησία και αξιολογεί και τη γνώριση των αρμοδιοτήτων τους και των, και τις επικοινωνιακές, επικοινωνιακές Υπενθυμίζω ότι πριν από την ακρόαση η υποψήφια επίτροπος έχει απαντήσει γραπτός ένα προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο και έχει διανεμηθεί το κείμενο αυτό σε όλες τις γλώσσες. Τέλος, παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν ε, είχε καμία αντίρρηση για την εξαγωγή αυτής της ακρόασης. Χαίρετε. Σας καλωσορίζω εδώ στην ακρόασή μας της υποψηφίας Επιτρόπου κυρίας Ντάλη, την οποία καλωσορίζουμε θερμά. Λοιπόν, ε, να σας παρουσιάσω τη διαδικασία της σημερινής μας συζήτησης. Πρώτα απ' όλα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ντάλη για 15 λεπτά για να κάνει μια εισαγωγική ομιλία για τις προτεραιότητές της. Κατόπιν θα έχουμε 25 ερωτήσεις από συναδέλφους σε δύο γύρους στον πρώτο γύρο επτά ερωτήσεων θα πάρουν το λόγο οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων και στο δεύτερο γύρο όπου θα πάρουν το λόγο 18 συνάδελφοι θα διανεμηθούν ε, μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων και θα πάρει το λόγο και ένας εκπρόσωπος των μη εγγεγραμμένων. Η συζήτηση θα γίνει με βάση τμήματα 5 λεπτών. Δηλαδή, ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση και κατόπιν ένα λεπτό στο ίδιο μέλος για μια συμπληρωματική ερώτηση και ένα λεπτό για την συμπληρωματική απάντηση. Σας παρακαλώ, ο χρόνος μας είναι αυστηρά προκαθορισμένος, θα είμαστε λοιπόν πολύ αυστηροί στην τήρησή του. Γι' αυτό έχω και το σφυράκι και θα το χρησιμοποιήσουμε δεν θα διστάσουμε. Σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας, ούτως ώστε όλα να διεξαχθούν ομαλά. Χθες είχαμε την πρώτη ακρόαση με τον ε, υποψήφιο επίτροπο κύριο Σμιτ και όλα πήγαν πολύ καλά. Παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι υπάρχει διερμηνία προς 23 γλώσσες ακριβώς αντανακλώντας τη γλωσσική πολυμορφία του σώματος. Όλοι οι ομιλητές μπορούν λοιπόν να μιλήσουν στη γλώσσα τους. Παρ' όλα αυτά, σας υπενθυμίζω ότι αυτά που θα πείτε θα πρέπει να μεταφραστούν. Σας παρακαλώ, όποια γλώσσα και αν χρησιμοποιήσετε, να μιλάτε με έναν ομαλό ρυθμό. Να έχετε πάντα υπόψη ότι οι ε, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να συμμεταφράσουν μεταφράσουν όσο καλύτερα γίνεται. Τέλος, η συζήτηση μεταδίδεται ζωντανά από το διαδίκτυο, το site του Κοινοβουλίου και θα έχετε δυνατότητα να δείτε και μια μαγνητοσκόπηση της συζήτησης στο ίδιο site του Κοινοβουλίου. Και τώρα ας ξεκινήσουμε να σας δώσουμε τον λόγο υποψήφια επίτροπε σας παρακαλώ να τηρήσετε τα 15 λεπτά που έχετε στη διάθεσή σας για την εισαγωγική σας ομιλία. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμοι ε, πρόεδροι, αξιότιμοι κύριοι ευρωβουλευτές, είναι σήμερα μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ ενώπιον σας σήμερα. Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα είχα την ευκαιρία να συζητήσω κάτι στο οποίο έχω αφιερώσει ολόκληρη την πολιτική μου ζωή, την ισότητα. Αφού ορίστηκα ως ε, ε, υποψήφια ώστε να προωθήσω αυτό το χαρτοφυλάκιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο Κοινοβούλιο εδώ οι, συζητή, τα, οι ιδέες συζητώνται από ένα μεγάλο φάσμα προοπτικών και είμαι πεπισμένη ότι αυτό που μας ενώνει είναι πολύ σπουδαιότερο από αυτά που μας χωρίζουν ή μας διχάζουν. Η ισότητα είναι ένας απεριόριστος πόρος Υπάρχει όντως αρκετή ισότητα για όλους και μπορούμε να τη στηρίξουμε. Από την άλλη πλευρά, οι διακρίσεις αποκλείουν, περιθωριοποιούν και οδηγούν μέλη της κοινωνίας μας το χείλο του γκρεμού. η διακρίσεις είναι μία άσκοπη πρακτική. Ε, ε, αποκλείει μέλη της κοινωνίας από την ευημερία, την πλήρωση και την ε, καλή ζωή. Ναι, βλάπτει το άτομα, τις μειονότητες, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. Γιατί αποσυνδέει τις ε, σχέσεις, μειώνει την εμπιστοσύνη και αλωτριώνει τους ανθρώπους. Η δημιουργία ενό ε, χαρτοφυλακίου αποκλειστικά για την ισότητα είναι ένα πολύ τολμηρό, μια τολμηρή δήλωση από πλευρά τη Προέδρου Φόντερ Λάιεν όσον αφορά την προώθηση τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ελευθεριών τη δημοκρατία καθώ και του κράτου δικαίου που ενισχύονται και προτάσσονται όσο στόχοι. Μια Ευρώπη άνευ διακρίσεων. Αυτή η εξέλιξη ακολουθεί τη δημοσίευση των πρώτων πολιτικών κατευθυντηρίων γραμμών που περιλαμβάνουν ένα ολόκληρο τμήμα για την ισότητα με σαφή μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν στη διάρκεια αυτής της θητείας και με τη δημιουργία της πρώτης επιτροπής με ισορροπία των φύλων. Η υποψήφια πρόεδρος έχει εκθέσει το όραμά τη και αν έχω εγώ τη στήριξή σας μετά από αυτή την ακρόαση είμαι έτοιμη να εργαστώ σκληρά με την ειδική ομάδα εργασίας για την ισότητα που δημιουργείται ε, γι' αυτό ακριβώς το σκοπό επιμονή μου βάσεως και αποτελείται από ανώτατους εκπροσώπους όλων των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της οποίας θα προεδρεύει ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής που είναι υπεύθυνο για τον πολιτικό συντονισμό. Και αυτό σε συνεργασία με το δικό μου επιτελείο, τις γενικές διευθύνσεις, την ε, θεματική, ε, τις θεματικές ομάδες υψηλού επίπεδου για την ισότητα των φύλων και την ε, καταστολή των διακρίσεων, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και την Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Επιπλέον, Σκοπεύω να συνεργαστώ σε διάλογο μαζί σας, ε, τους ευρωβουλευτές, καθώς και με τα κράτη-μέλη και την κοινωνία των πολιτών. Σκοπεύω να συνεργαστώ με όλους χωρίς να δαχτυλοδείχνουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να εξυψώσουμε τον τομέα αυτό τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός. Στη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε πολλούς ε, ε, σημών, ε, καθώς και με τις, ε, τα intergroup κατά των διακρίσεων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και με ε, δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών κατά των διακρίσεων τις τελευταίες εβδομάδες, έχω βρει ότι έχουμε πολλά κοινά στοιχεία. Συμφωνούμε ότι πρέπει να επιτείνουμε την αποφασιστικότητά μας υπέρ της ισότητας των φύλων, να επιτείνουμε τον αγώνα κατά της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων, καθώς και να προωθήσουμε την ισότητα επί τη βάση φύλου, ε, εθνοτικής προέλευσης, ηλικίας, ε, αναπηρίας, ε, θρησκείας, η πίστης και σεξουαλικού προσανατολισμού. Στις συζητήσεις που είχα, πολλοί εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τον προσανατολισμό αυτού του χαρτοφυλακίου επίσης και για τις ε, οριζόντιες και ε, κάθετες διαστάσεις του και μου ζήτησαν να δώσω σάρκα και οστά στο όραμά μου για το πώς ακριβώς όλα αυτά θα εφαρμοστούν. Η ισότητα πρέπει να ε, ισχύει για όλους και όλοι πρέπει να είμαστε μέρη αυτής της διαδικασίας ανάπτυξή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεχίσει να παίζει γετικό ρόλο παγκοσμίω σε αυτόν τον τομέα. Εγώ σε όλο μου το βίο έχω κάνει οτιδήποτε μπορούσα για να βελτιώσω τις ζωές των πολιτών. Μπήκα στην πολιτική, ίσως ε, όπως και πολλοί από εσά εδώ σε αυτήν την αίθουσα, όταν ήμουν φοιτήτρια 17 ετών, γεμάτη ενθουσιασμό, αφοσίωση και ιδεαλισμό. Με την πίστη ότι ασχολούμενοι, ακούγοντας, εξτρατεύοντας καθημερινά, θα μπορούσα να επιφέρω θετικές αλλαγές στην κοινωνία. Πολλά χρόνια αργότερα ξέρω πολύ καλά ότι αυτός ο αγώνας πόρο απέχει από το τέλος του. Αλλά έχω αποκομίσει ένα σημαντικό δίδαγμα, ότι οι πραγματικές αλλαγές είναι δυνατές μόνο αν εμείς οι πολιτικοί έχουμε το στένος να κάνουμε τις αλλαγές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Ο 21ος αιώνας οφείλει να είναι ο αιώνας ε, της ισότητας ε, των γυναικών. Ακριβώς πριν 40 χρόνια, το 1979, η Σιμών Βέιλ εξελέγει ως η πρώτη ε, γυναίκα πρόεδρος αυτού του κοινοβουλίου, ε, μιας από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές συνελεύσεις του κόσμου. Σήμερα, το 2019, χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να είναι σε όλες τις σφαίρες της ζωής τους μέσω μιας φιλόδοξης διαδικασίας ε, ένταξης του φύλου σε όλες τις πολιτικές τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών της όσο και των ε, σχετικών ε, αποτελεσμάτων τους. Ε, σήμερα, το 2019, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε την πεποίθησή μας και την εμπειρία, την ενέργεια που έχουμε για να φτιάξουμε δικαιότερες κοινωνίες στην Ένωση. Όπως είπε η πρόεδρος Φόντερ όσοι έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες θα πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να τις υλοποιήσουν. Και ξέρω πως είναι ένας ε, ανηφορικός αγώνας. Εγώ, ως Υπουργό Υπεύθυνο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις και την Ισότητα σε εθνικό επίπεδο, εργάστηκα σκληρά για να καταπολεμήσω τα κοινωνικά στερεότυπα, να καταθέσω νομοθετικές προτάσεις, να υιοθετήσουμε στρατηγικές και επίσης να στηρίξω, ε, μάλλον να, να αντισταθώ σε εκκλήσει ώστε να αμβληθούν τέτοιου είδου πρωτοβουλίες ισότητας. Ως Επίτροπος θα χρησιμοποιήσω παρόμοια προσέγγιση και θα δουλέψω με τα κράτη-μέλη ώστε να τους πείσω πως αυτές οι δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι σωστές. Διότι η πρόθεση της ένταξης και της ισότητας είναι ευρωπαϊκά ζητήματα όπως είναι και η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, η επίλυση των οικονομικών κρίσεων. Είναι ένας αγώνας που χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση και την πλήρη προσοχή μας. Επιτρέψτε μου τώρα να σας δώσω μερικά αριθμητικά στοιχεία, γιατί κάμια φορά οι αριθμοί μπορούν να πούν πολύ περισσότερο από ό,τι οι λέξεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 31% των γυναικών εργάζονται σε θέση μερικής απασχόλησης σε μεγάλο βαθμό γιατί φέρουν ε, τις περισσότερες ευθύνες της ανατροφής των παιδιών και της φροντίδας των ηλικιωμένων. Μία στις τρεις γυναίκες ε, φίσταται έμφυλη βία τουλάχιστον μία φορά στην ενήλικη ζωή της. Περισσότεροι από τους μισούς ε, μουσουλμάνους που αναζητούν ε, οικία υφίστανται διακρίσεις λόγω των ε, ονομάτων τους. Στο μικρού του επιθέτου το 80% των Ρωμά ζουν κάτω από το κατόφλι της στόχιας της ίδιας τους χώρας. 50% των πολιτών με αναπηρία δεν έχουν πρόσβαση στην εργασία και αποκλείονται. ηλικιωμένοι οι μεγαλύτερη ηλικία καλούνται κατά 39% λιγότερο σε συνεντεύξεις ε, για μια θέση εργασίας, ακόμα και όταν έχουν ακριβώς το ίδιο προφίλ και τα προσόντα με νεότερους. Δύο στους πέντε διεμφυλικούς ε, τρανς είναι κάθε χρόνο ε, θύματα βίας και σε τουλάχιστον 21 κράτη-μέλη γίνονται ιατρικές επεμβάσεις για να επιβάλλουν ένα φύλλο σε μεσοφιλικά παιδιά. Αυτή η χονδροειδής διάκριση ε, μπορεί να διευρύνεται όταν ε, υπάρχει ένα πρόσωπο που ανήκει σε διάφορες από αυτές τις ομάδες. Θα πρέπει να αναλάβουμε δράση και να ε, αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των αξιών που είναι τόσο προσφυλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιότιμα μέλη. Θα κάνω προσωπική μου μάχη, τη μάχη κατά των αποκλεισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα διστάσω να χρησιμοποιήσω κάθε εργαλείο για να προωθήσω την ισότητα και να ενισχύσω την προσήλωση της Ευρώπης στην ένταξη όλων και με κάθε μορφή της. Θα ήθελα να εστιάσω την εργασία μου κυρίως στα εξή τρία. Στην καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε είδους, στην συμπερίληψη και χειραφέτηση των γυναικών και στην προώθηση ισότητας και πλήρους συμμετοχής. Όλα αυτά ισχύουν για γυναίκες και άνδρες, για μειονότητες εθνοτικές και φιλετικές, θρησκευτικές σημεί, άτομα με αναπηρία, μεγαλύτερους και νεότερους σε ηλικία και ΛΟΑΤΚΙ. Ευθύς εξ αρχής μόλις αναλάβω θα ε, αναζητήσω τη βοήθεια και την υποστήριξη των συναδέλφων επιτρόπων για να προτείνουμε ό,τι χρειάζεται έτσι ώστε να προωθήσουμε την ε, ισότητα εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το σκοπό αυτό, μέσα στο πρώτο τρίμηνο από την ανάλυση των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συστήσω ομάδα δράσης Task Force για την ισότητα. Θα έχει ως εντολή ε, την περίπλοκη αποστολή της γρήγορης διατομεακής προσέγγισης για την ισότητα σε όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόθεσή μου είναι η Task Force να καταστεί επιχειρησιακή το δυνατότερο το γρηγορότερο δυνατό μάλλον, και να ε, είναι σωστά στελεχωμένη για να αντιμετωπίσει το τεράστιο αυτό έργο τη ένταξη τη ισότητα σε όλε τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, θα προτείνω μια νέα στρατηγική για το φύλλο με νέε νομοθετικέ προτάσει και εχμηρά μέτρα πολιτική. Έχει έρθει η ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις και τις δικές σας και της κοινωνίας των πολιτών μέσα στις πρώτες 100 ημέρες θα προτείνω νέα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τη διαφάνεια στις αμοιβέ. Είναι από τις βασικές μου προτεραιότητες κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Επίσης, θα επιμείνω στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό ε, χάσμα, έτσι ώστε να μην ορίζει το ποιοι είμαστε, το πόσο θα πληρωθούμε. Ή αν θα πληρωνόμαστε το ίδιο, αν θα έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες με κάποιους άλλους. Ως Επίτροπος για την Ισότητα θα παρακολουθώ ε, την πλήρη και σωστή εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη και από όλα τα κράτη-μέλη της οδηγίας ε, για την ισορροπία ιδιωτικού επαγγελματικού βίου. Δεν μπορώ να δεχτώ να φτάνει ακόμα τα 370 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως ε, η οικονομική απώλεια ε, λόγω ε, αυτού του προβλήματος ε, στην αγορά εργασίας. Θέλω να επιτύχει αυτή η υπόθεση της ισορροπίας ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί με τα κράτη-μέλη τα στερεότυπα του φύλου. Να βελτιωθούν οι δομές και οι υποδομές για την φύλαξη και υποδοχή παιδιών. Επίσης, δεν θέλουμε αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρίες και σε κάθε νομοθεσία θα πρέπει να ε, δίνεται προσοχή για την αναπηρία. Το 2020 αναμένεται ότι ένας στους έξι Ευρωπαίους πολίτες θα έχει κάποιο βαθμό αναπηρία. Εδώ λοιπόν ε, θα δώσω προτεραιότητα στην εφαρμογή της σύμβασης του ΙΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Και επίσης υπάρχει μια στρατηγική η οποία αυτόν τον καιρό αξιολογείται. Θα ήθελα να καθίσω μαζί σας αγαπητοί βουλευτές και να συζητήσουμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε και να προχωρήσει αυτό το πλαίσιο πολιτικής. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να προχωρήσει η βασική νομοθεσία στον τομέα της ισότητας. Ω υπουργό συμμετείχα σε ατέρμονες συζητήσει στο Συμβούλιο για προτάσει που παρέμειναν σε εμπλοκή για υπερβολή μεγάλο διάστημα, Όπω η οδηγία κατά των διακρίσεων που προτάθηκε πριν από 11 και πλέον έτη, ή οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια από το 2012 για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, του Συμβουλίου της Ευρώπης που ανάγεται στο 2016. Όλα αυτά πώς μπορούμε να τα εξηγήσουμε στου πολίτες μας. Στο πλαίσιο αυτό Εάν δεν καταφέρω ε, να ε, ρίξω τα ε, εμπόδια που υπάρχουν ακόμα και τους φραγμούς και αν δεν πείσω τα κράτη-μέλη που ακόμα έχουν επιφυλάξεις, δεν θα διστάσω να προχωρήσω στην εξέβραση νέων λύσεων και να προτείνω νέα νομοθεσία. Αυτό το οφείλουμε στους πολίτες μας, αυτή την πολιτική αλλά και το μετασχηματισμό τους πολίτες που αγωνίζονται για να τα βγάλουν πέρα και που υποφέρουν από τη βία θα πρέπει οι γυναίκες να ενισχυθούν, να χειραφετηθούν και ε, ε, τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες να υποφελούνται εξίσου. Ο δρόμος για να προχωρήσουμε είναι να ενταχθεί η ισότητα σε όλους τους τομείς πολιτικής. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και να περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις από πλευρά των συντονιστών των πολιτικών ομάδων. Και να δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στην κυρία Frances Fitzgerald. Έχετε αποδείξει ως υπουργό στη Μάλτα ότι έχετε κάνει πολλά για την ισότητα και εντυπωσιάστηκα όταν σας γνώρισα. Η δέσμευσή σας και οι ικανότητές σας επίσης είναι γνωστά. Ωστόσο, ως πρώτη ομιλήτρια δεν θα μπορούσα παρά να θέσω το εξή θέμα. Το Κοινοβούλιο ανησυχεί για την κατάσταση στη Μάλτα όσον αφορά τον απολογισμό και τις αξίες της κυβέρνησής σας σε σχέση με δύο συγκεκριμένα θέματα. Πρώτον, η δολοφονία της δημοσιογράφου που έκανε έρευνες Δάφνη Καρουάνα Καλίτσια. Η οικογένειά της ε, μας παρακολουθεί, πιστεύω σήμερα. Είστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο που έχει γίνει για τη διαλεύκανση και την ε, Δημόσια Εξεταστική Επιτροπή. Πώς θα επιχειρήσετε να προστατεύσετε δημοσιογράφους για να μην γίνουν τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα στο μέλλον. Είναι μια ευκαιρία να διευκρινίσετε τις απόψεις για το θέμα αυτό. <coughs> Δεύτερον, τα έργα του Παναμά, όπου ένας ε, συνάδελφός σας στην κυβέρνηση, ένας υπουργό ε, αναφέρθηκε. Συμφωνείτε με αυτά που έκανε αυτός ο υπουργό. Τι διδάγματα έχετε εξαγάγει και πώς θα τα εφαρμόσετε ως επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και ευχαριστώ για τα καλά λόγια που, είπαμε, που είπατε για μένα. Και εγώ πρέπει να πω ότι εκτιμώ την ε, δική σας στάση. Αναφερθήκατε σε αυτό το τραγικό έγκλημα, τη δολοφονία μιας γυναίκας της δημοσιογράφου Ντάφνη Καρουάνα Γκαλίτσια. Πρέπει να πω ότι οι εξαιρετικές καταστάσεις απαιτούν εξαιρετικά μέτρα. Θελήσαμε να εμπλακούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, όπως η Europol και το NFI και διεθνείς θεσμοί, όπως το FBI. Θυμάμαι ότι και εγώ είπα ότι το NFI θα έπρεπε να εμπλακεί στην έρευνα αυτή, γιατί τους γνώριζα. Εγώ είχα διοργανώσει αποστολές του NFI στη Μάλτα για να εκπαιδεύσουν τους δικούς μας αστυνομικούς σε θέματα ερευνών. Και πρέπει να πω ότι υπήρξε ουσιώδης πρόοδος. Σε 50 μέρες συνελήφθησαν τρία άτομα εντός 50 ημερών και τους απευθύνθηκε η κατηγορία, τους απαγγέλθηκε η κατηγορία. Συνεχίζεται, όπως ξέρετε, η έρευνα για το έγκλημα αυτό και για αυτά τα οποία είπατε. Βεβαίως θα κάνω ό,τι μπορώ τους ώστε ο τύπος να μπορεί να ασκεί ελεύθερα τα καθήκοντά του χωρίς φόβο και χωρίς πιέσεις. Με ρωτήσατε αν συμφωνώ με τις ενέργειες ε, του Υπουργού. Όχι, δεν συμφωνώ. Εγώ θα είχα δράσει εντελώ διαφορετικά. Σε όλη μου την πολιτική σταδιοδρομία αγωνίστηκα για σωστή διακυβέρνηση, για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία. Και ως υπουργό έκανα προσπάθειες, πρόθεσα για να υπάρξει η δημιουργία της θέσης του Επιτρόπου για την σωστή δημόσια ε, διαχείριση των υποθέσεων. Συγγνώμη, σας υπενθυμίζω ότι αυτό είναι ο κανόνας. Μία, ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση. Ένα λεπτό στην συμπληρωματική ερώτηση, ένα λεπτό για συμπληρωματική απάντηση. Και πρέπει να είμαστε αυστηροί από την αρχή, ώστε όλα τα μέλη να γνωρίζουν ότι πρέπει να σέβονται τους κανόνες. Και βεβαίως και εσείς κύριε υποψήφια επιτροπή. Παρακαλώ. Οπότε να δώσω το λόγο και πάλι στην κυρία Φιτζέρολ τη συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Τα θέματα του κράτου δικαίου και η ελευθερία του τύπου και η ανεξαρτησία δικαιοσύνη είναι κεντρική σημασία σε οποιαδήποτε στρατηγική ισότητα των φίλων. Γι' αυτό έθεσα αυτή την ερώτηση. Λόγω των ανησυχιών για τα θέματα αυτά από διάφορε ομάδε του Κοινοβουλίου, αλλά για θέματα στρατηγική για την ισότητα των φίλων που θέλετε να εκπονήσετε. Σα παρακαλώ, πέστε μα περισσότερε λεπτομέρειε. Σε τι θα βασιστεί αυτή η στρατηγική, ποια μεθοδολογία θα ακολουθήσετε τι διαβουλεύσεις θα κάνετε με ΜΚΙΟ και τι χρονοδιάγραμμα έχετε υπόψη σας. Ευχαριστώ. Ξέρετε, έχουμε πολλά να κάνουμε, αλλά αυτή η στρατηγική για την ισότητα των φύλων θα ασχοληθεί με τη διαφάνεια στις αμοιβέ, ε, τη συμμετοχή και των δύο φύλων την ψαλίδα στις συντάξεις και τους μισθούς, ε, την βία κατά των γυναικών και τα στερεότυπα φίλων ή φίλου. Γιατί δεν αρκεί η νομοθεσία. Πρέπει να αλλάξουν και οι νοοτροπίες. Θα ασχοληθώ λοιπόν συγκεκριμένα με τα θέματα αυτά των ε, στερεοτύπων των προκαταλήψεων λόγω φύλου. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε κατά τη διάρκεια της θητείας για να επιτύχουμε την ισότητα φύλων. Θα είναι αυτά τα τμήματα της στρατηγικής μου. Η κυρία Ρέγνερ. Τώρα ερωτώ εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων ε, αξίζει κάτι πάνω από μια συμπληρωματική ερώτηση. Ε, λοιπόν, κυρία υποψήφια επίτροπε, τονίσατε ότι είναι προτεραιότητά σας η στρατηγική αυτή ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων. Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι θα υπάρχει ακριβώς δεσμευτική ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέσα και τα εργαλεία έτσι ώστε να εφαρμόζεται. Σκέφτεστε μέτρα ελέγχου, συγκριτική αξιολόγηση, κυρώσεις. Και τι θα γίνει με την οδηγία για τις γυναίκε στα διοικητικά συμβούλια, θα είναι τμήμα τη στρατηγικής αυτή. Ποιε είναι οι συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλάβετε για να σπάσει αυτή η απεμπλοκή, αυτή η αφόρητη κατάσταση στο Συμβούλιο και να ε, τηρήσουμε αυτό το στόχο του 40% δεσμευτικό. Τι θα κάνετε γι' αυτό, η κυρία Επίτροπος. Βεβαίως, θα εργαστώ προς την κατεύθυνση της απεμπλοκής της οδηγίας σχετικά με τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Είναι όνειδος η κατάσταση αυτή τόσο καιρό. Θυμάμαι, από τις πρώτες μου δράσεις ως υπουργό ήταν να αλλάξω τη θέση της χώρας μου ε, σε αυτό ακριβώς το θέμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η προθυμία μου όσο και η δέσμευσή μου προς την κατεύθυνση αυτή με την οδηγία σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια για να γίνει πραγματικότητα. Φυσικά, λοιπόν, θα συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη και θα τα πείσω για την προστιθέμενη αξία αυτής της οδηγίας και ότι θα πρέπει να απεμπλακεί στο Συμβούλιο. Βεβαίως, με ρωτήσατε και για την στρατηγική ισότητα των φύλων εξίσου σημαντική για όλους μας. Θα εκδοθεί προσεχώς και φυσικά θα λάβω υπόψη τη διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους. Θα έχω τις απαραίτητες επαφές και θα βρούμε τα απαραίτητα εργαλεία έτσι ώστε σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές να εντάσσεται η διάσταση του φύλου αλλά να αναβαθμιστεί. Ξέρετε ότι αυτό είναι και ε, το έργο της ομάδας εργασίας Task Force ε, που είναι εγκάρσια σε όλες τις γενικές διευθύνσεις για να εξασφαλίζει ότι υλοποιείται πραγματικά αυτή η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Συμπληρωματική ερώτηση για ένα λεπτό. κυρία Ρέγνερ. Επανέρχομαι στην οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Θα προτείνετε κάποιες αλλαγές στο κείμενο το οποίο εκρεμεί τόσα πολλά χρόνια όπως αναφέρατε και ε, σχεδιάζετε άλλα μέτρα για να εξασφαλίσετε ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στις ε, ευρωπαϊκές υψηλές ε, θέσεις. Νομίζω ότι είναι ισορροπημένη η πρόταση. Θα συναντηθώ με όλους τους υπουργούς που έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για την πρόταση αυτή και θα πιέσω για να βρεθεί μια κοινή θέση στο Συμβούλιο. Thank Μάλιστα. Και τώρα ξανά το λόγο ως πρόεδρος και θα δώσω το λόγο στον επόμενό μας ε, ομιλητή εξ ονόματος της ομάδας Renew, η κυρία Ιρένα Καλημέρα σας. Όπως είπατε σωστά πριν από λίγο, πριν από ακριβώς 40 χρόνια εξελέγει η Σιμών Βέγη, πρώτη πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Είχε αφιερώσει τη σταδιοδρομία της στο να υπερασπίσει την δύναμη των γυναικών και έτσι έγινε για όλους μας ε, ίνδαλμα. Όμως ε, αυτές οι κατακτήσεις απειλούνται, όπως ας πούμε ε, εκτός Ευρώπης αλλά και στην Ευρώπη όπου 15 εκατομμύρια γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε νόμιμη ε, άμβλωση. Αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο. Ε, οι αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του σεβασμού, της ισότητας, όπως και το άρθρο, το σχετικό της, ονομα... της ε, τη Συνθήκης της Ένωσης, το ορίζει και όπως το δικό σας χαρτοφλάκιο το αποδεικνύει. Μπορείτε εσείς να μας πείτε ποιες θα είναι τώρα οι δικές σας συγκεκριμένες δράσεις ώστε να προωθηθούν τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, υπό ποια ε, με Πώς σκοπεύετε να συνεργαστείτε με τον Επίτροπο Αρμόδιο για την Υγεία για να εξασφαλίσετε τα αναπαραγωγικά δικαιώματα μέσα στο πλαίσιο μιας μελλοντική ευρωπαϊκής πολιτικής για την υγεία. Όπως σωστά είπατε, τα γυναικεία δικαιώματα τα δικαιώματα της γυναίκας μάλλον είναι ανθρώπινα δικαιώματα και εγώ είμαι βαθιά πεπισμένη φεμινίστρια και έχετε τον λόγο μου ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν ώστε να προστατευθούν τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Ε, νομίζω πως ε, θα πρέπει να ε, τεθούν εντός των ε, ευρωπαϊκών πολιτικών και αυτές, αυτά τα δικαιώματα και βεβαίως θα επιμείνω σε κάθε βήμα όπου μπορεί να ε, προσκρούσω σε αντιστάσεις. Πιστεύω όμως ότι όταν κανείς ε, ε, επιμένει στις αρχές του βρίσκει συμμάχους που να είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν. Πρέπει επίσης να ανταποκριθούμε στους βιώσιμους στόχους του ΟΗΕ για την υγεία, υγεία και για την καθολική πρόσβαση σε σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία υγεία, ε, οικογενειακό προγραμματισμό και ε, όλα τις σχετικές προβλέψεις και έχετε το λόγο μου είναι μια εγγύηση ότι τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα θα είναι μέσα σε αυτήν την ε, προσπάθειά μου άνευ εξαιρέσεως. Μάλιστα, ευχαριστώ. Έχετε επερώτηση. Ναι, μάλιστα. Όλες αυτές οι επιθέσεις στην ουσία είναι επιθέσεις κατά της ισότητας των φύλων. Το δικαίωμα να αγαπάμε όποιον θέλουμε και να ζούμε τη ζωή μας όποιον θέλουμε, όπως θέλουμε. Ε, τι ενέργειες εσείς θα κάνετε ώστε να αναχαιτήσετε τις επιθέσεις κατά της ισότητας των φύλων και της ελευθερίας. Αυτό που θα κάνουμε είναι να επιμείνουμε και με τη δουλειά μας ε, θα πρέπει να αναχαιτήσουμε αυτή την αντίσταση, να αντιπαρατεθούμε ε, μένοντας ισχυροί και αγωνιζόμενοι. Και όπως είπα και πριν, βρίσκουμε συμμάχους για να οικοδομήσουμε συμμαχίες των προθήμων και να επιμείνουμε. Να μην εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες. Ναι, συμβαίνουν τέτοια πράγματα γύρω μας, αλλά πρέπει να είμαστε εμείς ισχυροί και να τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ για τους πράσινους τώρα. Η κυρία Άλις Μπα Κιούνκε. Ευχαριστώ κυρία Ντάλια. Για να έχουμε πραγματική ισότητα των φίλων πρέπει να μας σε όλους τους τομείς πολιτικής. Μέχρι τώρα, συγκεκριμένε συγκεκριμένες μορφές διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι μουσουλμάνες και οι μαύρες γυναίκες, ε, άτομα λοάδικοι, οι γυναίκες με αναπηρίες, οι μετανάστριες, οι γυναίκες από διάφορε μειονότητες δεν έχουν αντιμετωπιστεί σωστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των πολιτικών ισότητας. Είναι θετικό ότι για πρώτη φορά θα έχουμε μία επίτροπο για θέματα ισότητα. Ωστόσο, η ισότητα μεταξύ των διαφόρων φυλών, φυλετική ισότητα, δεν αναφέρεται στις αρμοδιότητές σας. Είπατε ότι θέλετε να ξεπεράστε το αδιέξοδο για να εγκριθεί αυτή η οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων. Κύριε Αντάλη, πώς ε, θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να δημιουργήσετε την ε, πολιτική συμμαχιών για να ξεπεράσετε αυτό το αδιέξοδο στο Συμβούλιο. Τι συγκεκριμένε δράσει θα αναλάβετε. Και αν δεν μπορέσετε να ξεπεράσετε το αδιέξοδο για αυτή την οδηγία, θα προτείνετε μια νέα οδηγία. Επίση, δεσμεύεστε να υπάρχει οριζόντια προσέγγιση παντού, ώστε να υπάρχει πλήρης προστασία κατά των διακρίσεων ε, για οποιονδήποτε λόγο. Παρακαλώ. Η οριζόντια οδηγία, σε αυτήν αναφερθήκατε. Ναι, αναφέρθηκα στην οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων. Πρώτα απ' όλα, θα περιμένω να δω τι θα γίνει στη συνάντηση ΕΠΣΚΟ στις 24 Οκτωβρίου. όπου θα συζητηθεί το θέμα αυτής της οδηγίας κατά των διακρίσεων και κατόπιν θα δω τι θα κάνω. Αλλά η βούλησή μου είναι να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο για αυτή την οδηγία. Γιατί όπως σωστά είπατε, υπάρχουν ακόμη πολλές διακρίσεις και η αντιμετώπιση τους πέρα από το τομέα της απασχόλησης στην Ένωση δεν είναι κάτι το προφανές. Φυσικά είναι μεγάλη πρόκληση γιατί Απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο. Αλλά θα το συζητήσω με όλους τους υπουργούς. Αλλά πρέπει γρήγορα να προχωρήσει το θέμα αυτό. Επίσης, είναι καλό που έχουμε ομάδες υψηλού επίπεδου που κάνουν πολλή δουλειά. Και είναι καλό αυτό. Και υπάρχει και η χάρτα για την ισότητα ουσιώδης. Αλλά θα συνεχίσω τις προσπάθειές μου για να υπερβούμε το αδιέξοδο για αυτήν την οδηγία. Κυρία Κιούνκε, για να υπάρξει στήριξη για μια νέα οδηγία που να τα περιλαμβάνει όλα, θα χρειαστείτε επίσης και στήριξη από άλλους επιτρόπους. Για παράδειγμα τον αντιπρόεδρό σας, τον κύριο Σχοινά, που έχει ως αρμοδιότητα την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και τη στήριξη της κυρίας Φόντερ της ίδιας. Όπως είπατε, θέλει να δημιουργήσει μια ειδική ομάδα, task force, για αυτό το θέμα. Πώς θα συνεργαστείτε με αυτήν την ειδική ομάδα για να αυξήθει η στήριξη στις ιδέες σας. Ναι, σωστά είπατε. Πρέπει να συνεργαστώ με τον Αντιπρόεδρο κύριο Σχοινά. Συμφωνούμε και οι δύο ότι η ισότητα είναι τμήμα του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Συμφωνούμε από αυτό. Και η πρόεδρος Φόντε έθεσε ακριβώς την ισότητα τη θέτει μάλλον, σε τόσο υψηλό επίπεδο που δημιούργησε μία επίτροπο για αυτό το θέμα. Και δημιούργησε και αυτήν την ειδική ομάδα που θα είναι υψηλού επίπεδου. Με υψηλό επίπεδο προσώπου από όλες τις γενικές διευθύνσεις. Αυτό είναι σαφής απόδειξη ότι θέλουμε να προχωρήσει το θέμα αυτό και θα προχωρήσει. Κυρία Κριστίνα Άντερσον από την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας καλύτερα κυρία Τάλη. Προηγουμένως τονίσατε ότι θέλετε να αγωνιστείτε έτσι ώστε να μπορούν να αποφασίζουν ελεύθερα όλοι οι άνθρωποι σε ποιο φύλλο θεωρούν ότι ανήκουν. Στις Ηνωμένε Πολιτείε. Συγγνώμη, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά δεν σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Παρακαλώ, μήπως μπορείτε να περιμένετε λίγο να επιβραδύνετε και να ξαναρχίσετε την ερώτησή σας. Αξιότιμη κυρία Ντάλη, μια στιγμή. Please, one little moment. Two. So, one little moment we instruct. Μια στιγμή. So, could you please... Λοιπόν, ε, σας παρακαλώ ε, να επαναλάβετε. Αξιότιμη κυρία Ντάλη, προηγουμένως τονίσατε ότι θα αγωνιστείτε έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα το φύλλο στο οποίο θεωρούν ότι ανήκουν. Στις Ηνωμένε Πολιτείε, σε ορισμένες πολιτείε ήδη, υπάρχει εξή πρακτική. Κάποιοι άνθρωποι ε, μπορούν να αλλάξουν φύλλο ε, επειδή το επιθυμούν οι ίδιοι, το ζητούν οι ίδιοι. Ε, πέρα από κάποιες εγχειρήσεις ή κάποιες γνωματεύσεις ε, αρμοδίων αρχών και μετά είναι κάποιοι υποχρεωμένοι να το δέχονται. Αυτό το θεωρείται σκόπιμο, πρακτική και ως επίτροπος θα συνηγορούσατε υπέρ ενός τόσο ευραίος έτσι, εννοούμενου δικαιώματος στην αυτοδιάθεση και στον αυτοπροσδιορισμό ελπίζω να ακούσατε τη διερμηνία, κυρία υποψήφια επίτροπε. Μάλιστα. Συμφωνώ με την νομοθεσία στην οποία αναφέρεστε. Ε, και στη χώρα μου, εγώ προχώρησα ε, σε αυτή την νομοθεσία. Εγώ την εισήγαγα στη Μάλτα. Η νομοθεσία αυτή εγκρίθηκε στη χώρα μου μετά από συναντήσεις που είχα πριν την προτείνω και από ανθρώπους που άκουσα τις ιστορίες τους, τη μαρτυρία τους. Συναντήθηκα με οικογένειες που είχαν διεμφυλικά, μεσοφιλικά παιδιά, transgender και intersex, στα αγγλικά οι όροι, και μου ανέφεραν, μου διηγήθηκαν τα δεινά και τον πόνο και τα όσα τραβούσαν οι οικογένειες αυτές. οι διεμφυλικοί, οι τρανς, δεν θέλουν να κάνουν εγχείρηση ε, προς διορισμού του φίλου, η αλλαγή φίλου, αλλά ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους και δεν ήθελαν να βγουν έξω, γιατί το όνομα που είχαν στα χαρτιά τους δεν αντιστοιχούσε με το πρόσωπο που ήδη έβλεπαν στον καθρέφτη και έχω στο μυαλό μου την θλιβερή ιστορία ενός κοριτσιού που αυτοκτόνησε γιατί δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι, γιατί τρεπότανε. Επειδή τα χαρτιά της, η ταυτότητά της, το διαβατήριό της, ο έλεγχος του σχολείου είχαν ένα όνομα αγοριού επάνω, αλλά η ίδια αισθανόταν κορίτσι, γυναίκα. Και όταν την έβλεπες, έβλεπες ένα κορίτσι όταν είσαι αντιμέτωπη με τέτοιες καταστάσεις, πώς είναι δυνατόν να μην προχωρήσει σε νομοθεσία, έτσι ώστε να βελτιώνονται οι ζωές των ανθρώπων αυτών, έτσι ώστε οι οικογένειες να μπορούν να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής καν. Θα μπορούσα να σας μιλήσω επίσης ε, από τη, ε, για την εμπειρία μου με μεσοφιλικά άτομα, intersex, που επίσης αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. ξέρω ότι το κοινοβούλιο σας έχει εγκρίνει σχετικά ψηφίσματα για τους μεσοφιλικούς και ως νομοθέτες και πολιτικοί νομίζω ότι γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να βελτιώνουμε τη ζωή των ανθρώπων. So, Uh, it's Συγγνώμη, αλλά η δουλειά μου είναι να σας κόβω το λόγο. Ε, έχουμε υπερώτηση ε, συμπραγματική από την κυρία Άντερσον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για την απάντηση. Ωστόσο, σε αυτή την πρακτική που να μπορεί κανείς κάθε τόσο να αλλάζει φίλο, βλέπω ένα μεγάλο κίνδυνο. Ε, ε, κάνουμε τόσες προσπάθειες για να σπάσουν ε, οι διακρίσεις κατά των γυναικών και τώρα αυτό πάει να γυρίσει ανάποδα με αυτές τις πρακτικές. Ας πούμε όταν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του γυναίκα και είναι άνδρας θα μπορεί να συμμετέχει στο γυναικείο αθλητισμό και αυτό είναι εις βάρος των γυναικών. Ή ας πούμε στα διοικητικά συμβούλια μπορεί κάποιο άνδρα να αλλάξει φίλο και να τον πάρουν στο διοικητικό συμβούλιο επειδή είναι γυναίκα για να τηρηθεί η ποσόστοση. Οι διακρίσει κατά των γυναικών πώς θα έρθουν όταν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να δηλώνει ότι αλλάζω φίλο και τώρα ανήκω στο τάδε φίλο. Και θα είναι και πολύ χειρότερα από ό,τι στο παρελθόν φοβάμαι. Όχι απλώς δεν θα έρθουν οι διακρίσεις. Η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ. αυτή η αλλαγή φύλου, η ταυτότητα του φύλου, δεν είναι ένας περίπατος στο πάρκο. Δεν βγαίνεις για βόλτα. It's not Δεν είναι κάτι που κάνει κάποιος έτσι αψήφιστα για να μπει σε ένα διοικητικό συμβούλιο ή να τρέξει σε ένα στίβο. Γεννιέσαι με αυτό. Αυτό σε βρίσκει. Δεν το βρίσκεις εσύ. Κάνει τη ζωή σου και τη ε, ζωή τη οικογένεια σου πολύ ε, θλιβερή, πολύ σκληρή. Και είμαι σίγουρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν τέτοιε περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρετε. Και σας παρακαλώ, α σεβόμαστε λίγο του ανθρώπους που έχουν ανάγκη το σεβασμό μας. Ε, που μας χρειάζονται εμάς για να τους βοηθήσουμε. Να κατανοήσουμε τις καταστάσεις που ζουν. Να μπούμε στο πετσί τους, στα παπούτσια τους όπως λέμε στα αγγλικά και να κάνουμε μερικά βήματα με τα δικά τους παπούτσια για να κατανοήσουμε τη ζωή που ζουν και την πραγματικότητα που ζουν. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βοηθάμε τους ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, που αν δεν κάνουμε εμείς κάτι θα ζουν μια άθλια ζωή και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Thank you. Uh, the next question goes to the ECR uh, Επόμενη ερώτηση της κυρίας Βυ Βυζνιέσκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς μιλάτε διαρκώς για σεβασμό και θα περίμενε κανείς ότι οι επιτροπές που συνεδριάζουν εδώ θα έπρεπε να σέβονται τις απόψεις όλων μας και του προηγούμενου ομιλητή, γιατί και αυτή είναι μια μορφή διακρίσεων. Εσείς, Επίτροπε, εκπροσωπείτε μια χώρα της οποίας η νομοθεσία προβλέπει την απαγόρευση των αμβλώσεων. Στη συνθήκη Οι σχετικές διατάξεις και η νομοθεσία των κρατών μελών για οικογενειακά θέματα συμπεριλαμβανομένης της ε, άμβλωσης θα πρέπει να τηρούνται. Ωστόσο, τα ζητήματα αυτά τώρα συζητώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ασκούνται πιέσεις ώστε να ρυθμιστούν αυτά τα θέματα. Εσείς μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι θα σεβαστείτε τις συνθήκες, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αναπτύξουν τις νομοθεσίες τους χωρίς να τους ασκείτε καμία πίεση. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα αξιών και υγείας. Το άλλο θέμα είναι ο ακροτηριασμός γεννητικών οργάνων. 200.000 γυναίκες επηρεάζονται από αυτό το πρόβλημα. Επίσης υπάρχει και το θέμα των καταναγκαστικών γάμων που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έχετε να σχολιάσετε γι' αυτό. Παρακαλώ, κυρία υποψήφια επίτροπε. Yes, Μάλιστα. Όπως είπατε, η άμβλωση είναι αρμοδιότητα του των κρατών μελών. Και βεβαίως πάντοτε ε, θα σέβομαι τις συνθήκες. Και έχετε δίκιο για τον ακροτηριασμό των ε, γυναικείων γεννητικών οργάνων που είναι μια άλλη φρικτή πληγή αποτέλεσμα της ε, πατριαρχίας κάτι για το οποίο βεβαίως πρέπει να δουλέψουμε και πέρα από δράσεις και ίσως και σχετική νομοθεσία, νομίζω πως θα πρέπει να δούμε την καθημερινότητα που ζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και πώς μπορεί να επηρεαστούν. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα όπου ένα κορίτσι πρόσφυγας παρακολουθούσε το σχολείο και ξαφνικά σταματάει να πηγαίνει στο σχολείο. Ξανάρχεται μετά από δύο εβδομάδες αφού πιθανότατα τις έχουν κάνει ε, ακροτηριασμό. Πέρα από τα όσα μπορούμε να κάνουμε ως Ένωση, θα πρέπει να επαγρυπνούμε, πιστεύω, ως άνθρωποι στις κοινωνίες μας ώστε να προσέχουμε μήπως αντιληφθούμε τέτοιου είδους πράγματα, καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και το ίδιο και για τους αναγκαστικούς γάμους. Βεβαίως πολλά πρέπει να κάνουμε. Όμως το πρώτο που πραγματικά πρέπει να κάνουμε ο καθένας από μας είναι να νοιαστούμε για τους, ε, ε, τις κοινωνίες μας και να παρατηρούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Γιατί μπορεί να υπάρχουν νομοθεσίες, αλλά κάποιες φορές γίνονται και πράγματα τα οποία δεν τα αντιλαμβανόμαστε, δεν τα καταλαβαίνουμε. Ενώ όταν επαχρυπνάει, επαχρυπνά, παρατηρεί, ε, ρωτάει τι συμβαίνει, καταλαβαίνει πως συνεχίζουν να γίνονται τέτοια πράγματα. Μάλιστα, ευχαριστώ. 30 δευτερόλεπτα έχετε για την ερώτησή σας, γιατί η πρώτη σας ερώτηση διήρκησε πολύ περισσότερο. Θα ήθελα να σχολιάσετε με περισσότερες λεπτομέρειες το θέμα των ε, σεξουαλικών στερεοτύπων. Το Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το πρόβλημα. Πιστεύετε ότι ο ρόλος της μητέρας και της συζύγου είναι επίσης ένα ε, στερεότυπο φίλου. Και μπορείτε να διευκρινίσετε πώς θα καταπολεμήσετε τους αναγκωστικούς γάμους που στην ουσία είναι υποθέσεις παιδοφιλίας. Ε, stereotyping. Ναι, τα στερεότυπα είναι πολύ σημαντικό θέμα και θα αντιμετωπιστεί στην στατικική μας περί Η χρήση στερεοτύπων είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο κόσμος βλέπει με συγκεκριμένο τρόπο τους υπολείπους, δηλαδή σε σχέση με το πώς ε, αναμένεται να συμπεριφέρονται ή να εργάζονται με συγκεκριμένο τρόπο. Είπατε μητέρα, σύζυγος. Ναι, Χαίρομαι πολύ για την οδηγία περί ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής, γιατί πολλές φορές οι γυναίκες είναι θύματα στερεοτύπων. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε τη συμβολή των ε, πατέρων ανδρών στις ε, ε, οικογένειες. Υπάρχει αυτό το στερεότυπο ότι η μητέρα είναι πάντοτε ε, εκείνη που προσφέρει τη φροντίδα 100% και ο πατέρας είναι εκείνος που εργάζεται εκτός του σπιτιού. Ναι, τα στερεότυπα λοιπόν είναι πολύ αρνητικά και είναι αυτά που μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιες ε, περιστάσεις όπου Πρέπει να αλλάξουμε, όπως είπαμε, πράγματα και να νομοθετήσουμε και με την οδηγία ε, ισορροπή, ε, ισορροπίας ε, μεταξύ εργασιακού και οικογενειακού βίου κάτι κάνουμε, ας πούμε, για τη δεκαήμερο πατρικής άδειας. Ναι, είναι κάτι πολύ θετικό, γιατί έτσι όντως διαπιστώνουμε ότι και οι μητέρες και οι πατέρες πρέπει να ασχοληθούν με το μεγάλωμα των παιδιών τους και έτσι να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ της εργασιακής και της προσωπικής ζωής. Γιατί τα στερεότυπα είναι πολύ αρνητικά πάντοτε και ένας λόγος για τον οποίο φτιάχνουμε νομοθεσίες και οδηγίες ακριβώς είναι τα στερεότυπα. Πρόσφατα ε, χάρηκα που είδα κάποια καινούργια παιδικά βιβλία όπου αντικατοπτρίζεται η οικογενειακή ζωή όπως αυτή συμβαίνει ανάμεσα στα διάφορα μέλη. Τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν με νέα μοντέλα οικογένειας τώρα. Υπάρχουν βιβλία όπου οι γυναίκες είναι επιστήμονες, είναι καλλιτέχνες και αυτό βοηθά να σπάσουν τα στερεότυπα, να δείξουμε πως και οι μητέρες μπορούν να είναι επιστήμονες, μπορούν να είναι καλλιτέχνες, όπως και οι πατέρες το ίδιο. Αλλάζουν τα πράγματα νομίζω, αλλά πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Αχ, συγγνώμη, ξέχασα το ρολόι. Απλώς σας άκουγα, ξέχασα να βάλω το χρονόμετρο. Αυτό το λεπτό λοιπόν φάνηκε να κρατάει πολύ ώρα. Εν πάση περιπτώσει, όμως ο χρόνος ε, τρέχει. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Επόμενη ερώτηση είναι από την ομάδα της ΚΟΕ και την κυρία Σάντρα Περέιρα. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας κυρία Επίτροπε σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς δημόσιους ε, παιδικούς σταθμούς και η ιδιωτική είναι πολύ ακριβή για τις οικογένειες. Ένα ιδιωτικό δίκτυο ε, ε, είναι αυτό το οποίο λειτουργεί λοιπόν και τελικά αναγκάζονται οι γυναίκες να, κυρίως να αφήνουν την απασχόλησή τους για να φροντίσουν τα παιδιά και αυτό έχει επιπτώσει για την σταδιοδρομία τους αλλά και για για την ε, ε, οικογένεια. Η δημιουργία παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών είναι πολύ σημαντική για ε, την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Σα ρωτώ λοιπόν ποια είναι η στρατηγική τη επόμενη ε, Επιτροπή για την επίτευξη των στόχων τη Βαρκελόνη, εάν δηλαδή θα δοθούν περισσότερα χρήματα για προγράμματα και μέσα, ώστε να στηριχθούν τα κρατημέλη στο να αναπτύξουν ένα δημόσιο δίκτυο ε, σταθμών και ε, παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών σύμφωνα με τις ανάγκες και να αντιστοιχούν και στα κριτήρια του ελλείμματος. Ευχαριστώ, κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Είναι πολύ ουσιώδες για να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή και των δύο γονιών στην αγορά εργασίας. Και έχω και ίδια πείρα από τη Μάλτα. όπου έχει εισαχθεί η δωρεάν ε, βρεφονιπιακή και παιδική φροντίδα για γονείς που εργάζονται ή ε, είναι φοιτητές. Και έτσι αυξήθηκε εκθετικά η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Έτσι διαπιστώσαμε λοιπόν ότι οι γυναίκες δεν μπορούσαν να εργαστούν αν έπρεπε να δαπανούν ε, πολύ μεγάλα ποσά για την ε, βρεφονιπιακή φροντίδα. Ναι, πρέπει να κάνουμε περισσότερα, να βρούμε τρόπο, ούτως ώστε να υπάρχει τουλάχιστον προσιτή βρεφονιπιακή φροντίδα. Αυτό θα βοηθήσει και την εφαρμογή της οδηγίας συνδυασμού προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Που ακριβώς αυτό επιδιώκει. Το συνδυασμό προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Και σε αυτό το τομέα Πρέπει να κάνουμε πολλά και οπωσδήποτε θα το προωθήσουν για να υπάρξουν και επαρκείς πόροι για να εφαρμόσουμε μέτρα ούτως ώστε να υπάρχει ε, σε προσιτή τιμή αυτή η φροντίδα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ για τη συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, ήθελα να διευκρινίσω κάτι περισσότερο σε σχέση με τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Κάποιες χώρες έχουν ε, παναχωρήσει, επισοδρομήσει τα τελευταία χρόνια. Εμείς όμως δεν θέλουμε να πάμε πίσω. Πώς μπορείτε να συμβάλλετε ώστε να συνεχιστούν οι πρόοδοι και να ε, ε, πείσετε τα κράτη-μέλη να λάβουν τα μέτρα που εγγυώνται αυτά τα δικαιώματα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά για τις γυναίκες στη διάρκεια της ζωής, να ενισχύσετε την προσφορά ε, υγειονομικής περίθαλψης για τη σεξουαλική και αναπαραγωγικά δικαιώματα, Πώς θα, μπορέσετε, πώς θα τους πείσετε να χρηματοδοτήσουν προγράμματα για την κατάρτιση ειδικευμένων ε, γυναικολόγων αλλά και νοσοκομιακού ε, προσωπικού ώστε να γνωρίζουν και να ενημερώνονται για τις πιο καινοτόμες πρακτικές και τεχνολογίες. Ναι, οπωσδήποτε πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, των Ηνωμένων Εθνών και όσον αφορά την υγεία των γυναικών. Να υπάρχει πρόσβαση για όλες τις γυναίκες στην ε, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και να υπάρχει κατάρτιση για θέματα οικογενείας και με, τον, ε, με την Επίτροπο για την Υγεία και τον Αντιπρόεδρο για την ε, Δημοκρατία και το Δημογραφικό θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε οι προσπάθειες αυτές να συνεχίσουν να στηρίζονται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε ολοκληρώνουμε τον πρώτο γύρο και πριν περάσουμε στο δεύτερο γύρο υπενθυμίζω σε όσους θα λάβουν τώρα το λόγο ότι το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους υποψηφίους με βάση των γενικών ικανοτήτων τους, τη δεσμευσή τους για την Ευρώπη, την προσωπική ανεξαρτησία και τη γνώση του προτινόμενου χαρτοφυλακείο τους και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Λοιπόν, τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Κάζα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντάλη, αναφέρθηκε ότι το Κοινοβούλιο έκανε την πρώτη ανάγνωση της οδηγίας για τον συνδυασμό προσωπικής και επαγγελματικής ζωής <clears throat> και θέλουμε να υπάρξει ισότητα και στο καταμερισμό των ε, οικογενειακών ευθυνών. Νομίζω ότι κάθε διάκριση πρέπει να αποφευχθεί. Τι θα κάνετε λοιπόν τόσο ώστε να διασφαλίσετε ότι θα εφαρμοστεί αυτή η οδηγία με ουσιώδη τρόπο. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Για όλη την εργασία του Κοινοβουλίου <clears throat> για τα θέματα αυτά για αυτήν την οδηγία. Όπως ξέρετε, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα τριών ετών για την εφαρμογή της. Εάν ε, επικυρωθώ ως επίτροπος θα βοηθήσω και τη χώρα μου και τα άλλα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία. Ξέρετε πόσο πιστεύω σε αυτή την οδηγία και έχω πραγματικά δεσμευθεί στην εφαρμογή της. Πραγματικά θα ήθελα να λειτουργήσει σωστά, να εφαρμοστεί σωστά. Μπορούμε να έχουμε ειδικέ συνεδριάσεις, σεμινάρια για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να καταλάβουν πώς θα την εφαρμόσουν. Τι σημαίνει η εφαρμογή αυτή. Και πιστεύω ότι χρειάζεται και περισσότερη ευαισθητοποίηση των ίδιων των εργαζομένων να κατανοήσουν περί πρόκειται. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο εδώ. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν την ευθύνη να εφαρμοστεί πλήρω η οδηγία. Να καταλάβουν ότι θα ωφεληθούν όλε οι οικογένειε από την εφαρμογή αυτή. Γιατί θεωρώ ότι θα βοηθήσει πολύ τι κοινωνίε μα η εφαρμογή τη. Για παράδειγμα, θα βοηθήσει να καταρρύψουμε τα στερεότυπα. νου δουλειά είναι η φροντίδα των παιδιών ή άλλες δουλειές του σπιτιού θα μας βοηθήσει όλους. Κάθε οικογένεια θα πρέπει να οργανώνει τις δουλειές του σπιτιού με τον βέλτιστο τρόπο. Και αυτή η οδηγία θα βοηθήσει τις οικογένειες να επιτύχουν αυτή τη σωστή κατανομή ρόλων. Να αξιοποιήσουν καλύτερα τον ελεύθερο χρόνο τους, τα μέλη της οικογένειας, για να φροντίσουν για τα παιδιά ή για ηλικιωμένους έτσι ώστε όλοι να έχουν χρόνο για να ασχοληθούν με την οικογένειά τους. Εάν λοιπόν με βεβαιώσετε ως Επίτροπο, θα κάνω ό,τι μπορώ να βοηθήσω τα κράτη-μέλη να εφαρμόσω αυτή την οδηγία. Παρακαλώ, συμπληρωματική ερώτηση. Τώρα κάτι άλλο. Όπως ήδη ακούσαμε, έχει να κάνει και με το κράτος δικαίου. Είσαστε υπουργό. Και όπως ξέρουμε από τα έγγραφα του Παναμά, κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί αμείβονταν 5.000 ευρώ την ημέρα για κάποιες δραστηριότητες. Τι θα κάνετε ως Επίτροπος, ούτως ώστε να μην γίνονται τέτοια πράγματα στο μέλλον. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένας νόμος για τους μεν και άλλος για τους δε. Κοιτάξτε. Στην σταδιοδρομία μου στην πολιτική μέχρι τούδε πάντα ασχολήθηκα με τη χρηστή διακυβέρνηση, την πρόθεση δηλαδή, το κράτος δικαίου και είμαι υπέρ των θεμελιωδών αξιών των κοινωνιών μας. Ε, εργάστηκα για να δημιουργηθεί η θέση του Επιτρόπου για την χρηστή διακυβέρνηση και τις σωστές προδιαγραφές στο δημόσιο βίο. Και ε, ένας πολιτικός ε, αποκαλύπτεται ότι έχει διαπράξει αδικήματα, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι υπόλογος για αυτά. Και εργάστηκα πολύ για να περάσει ο νόμος για τους καταγγέλτες, ο νόμος για τα πολιτικά κόμματα στη χώρα μου, όλες αυτές τις δραστηριότητες Νομίζω ότι αποδεικνύουν ότι η στάση μου και τα διαπιστευτήριά μου για αυτή τη θέση είναι γνωστά. Τώρα ήταν καλή πρόεδρος, τώρα θα ακούσετε την κακή πρόεδρο. Θα είμαι αμήλικτη με το χρόνο. Η κυρία Γουαρμίνη από Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ένα λεπτό για την ερώτησή σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γουαρμίνη. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, όπως γνωρίζετε, το μεικτό ορομίσιο των γυναικών είναι 16% χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών και στις συντάξεις αυτό φτάνει ακόμα και στο 36% διαφορά. Ξέρουμε ότι η καταπολέμηση των ανισοτήτων είναι ύψιστη ε, προτεραιότητα και από την πολιτιστική σκοπιά και για τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, αλλά και ποσοτικά. Γιατί στην πολιτική παίζουν ρόλο και τα μαθηματικά. Όταν οι γυναίκες κάνουν την ίδια δουλειά, στο ίδιο επίπεδο, στον ίδιο χώρο εργασίας, θα πρέπει να αμείβονται με τις ίδιες αμοιβέ, όπως και οι άνδρες. Καλωσορίζω πάρα πολύ αυτό που είπατε για τη διαφάνεια προς τις ε, αμοιβέ. Τι θα κάνετε όμως για να μειώσετε ακόμα και να εξαλείψετε αυτό το χάσμα που υπάρχει ε, από νομοθετικά μέτρα ερωτώ που ελπίζω όλοι ελπίζουμε ότι θα εφαρμόσετε. Η κυρία Επίτροπος, ευχαριστώ. Όπως είπατε, όντως είναι 16% η διαφορά μεσολογική ανδρών και γυναικών εάν με επιβεβαίωσατε ως Επίτροπο, αυτό που σκοπεύω να κάνω και μάλιστα τις πρώτες 100 ημέρες είναι να εργαστώ επί μίας προτάσεως για τη διαφάνεια ως προς τα μισθολογικά. Γιατί δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει αυτό το χάσμα, τη διαφορά και την ψαλίδα και ενδεχομένως και τελικά και των συντάξεων, αν δεν υπάρχει διαφάνεια στις αμοιβέ. Από εκεί θα περάσει ο δρόμος. Αυτό είναι το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε, έτσι ώστε να δούμε ακριβώς πού βρίσκονται αυτές οι διαφορές. Όπως γνωρίζετε, η εκλεγμένη πρόεδρος μου ανέθεσε ε, τις πρώτες 100 ημέρες να ε, καταρτήσω και να καταθέσω την πρόταση αυτή για τη διαφάνεια ως προς τις αμοιβέ, αλλά και ε, στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για τη διαφάνεια προς τις αμοιβέ και για μέτρα που θα εξασφαλίζουν την ίδια αμοιβή για την ίδια εργασία ε, στον ίδιο χώρο εργασίας. Γνωρίζουμε ότι αυτή η μισθολογική διαφορά ανακλάται και στη διαφορά στην τάξη. Αναφέρατε κι εσείς ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και 36%. Ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό, διότι οι γυναίκες, ακόμα και αν αρχίζουν ε, να εργάζονται, με τα ίδια προσόντα, με την ίδια εμπειρία, όπως και οι άνδρες, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, μπορεί να χρειαστεί να δουλεύουν με μικρότερο ωράριο και πληρώνουν λιγότερες εισφορές. Άλλες φορές δουλεύουν σε μερική, ε, δουλεύουν σε μερική απασχόληση. Και αυτό θα βοηθήσει και η άλλη οδηγία. Ε, ε, πληρώνουν λοιπόν λιγότερες φορές και στο τέλος της καριέρας τους έρχονται να διαπιστώσουν ότι όχι μόνο έβγαζαν λιγότερα χρήματα από τους άνδρες για την ίδια δουλειά, αλλά και η σύνταξή τους θα είναι μικρότερη. Γιατί έχουν καταβάλει λιγότερες ε, συνταξιδοτικές εισφορές. Λοιπόν, είναι πολλή δουλειά που μας περιμένει και η αφετηρία είναι αυτή για τη διαφάνεια. Η συμπληρωματική ερώτηση, ένα λεπτό παρακαλώ. Άρα, δύο πολύ ε, σύντομες ε, συμπληρωματικές ερωτήσεις. Πρώτον, προτίθεστε να συμπεριλάβετε και τους κοινωνικούς εταίρους σε αυτές τις ε, διαβουλεύσεις και σε κάποιες προκαταρκτικές συμφωνίες για την οδηγία για την ισότητα στις Και δεύτερον, προτίθεστε στα νομοθετικά μέτρα για τις αμοιβέ θα βάλετε και κάποιους δείκτες για να μπορείτε να παρακολουθείτε και να αξιολογείτε τον αντίκτυπο και τη σωστή εφαρμογή των νομοθετικών αυτών μέτρων. Φυσικά. Η κοινωνική εταίρη είναι πολύ σημαντική για μας και είναι τμήμα της διαβούλευσης και της πολιτικής αυτής, της συγκεκριμένης πρότασης. Έτσι εργάζομαι. Έχω διατελέσει υπουργός κοινωνικού διαλόγου και κοινωνικών ε, σχέσεων των κοινωνικών εταίρων μεταξύ τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Είναι ενεχόμενοι να συμμετέχουν όταν θέλεις να κάνεις κάτι που επηρεάζει κυρίως την απασχόληση και αφορά ε, τα θέματα αυτά φυσικά. Και επίσης θα έχουμε και μέτρα και δείκτες για να μετρούμε την απόδοση και τις επιδόσεις. Για να προχωρούμε βάσει αξιολογήσεων ε, αν χρειάζεται να αναθεωρούμε, να τροποποιούμε και να βελτιώνουμε. Μάξοβα, your question, one minute. Κυρία Μάξοβα, για ένα λεπτό. Ehm, Ευχαριστώ. Και εσείς στην ε, ε, εισαγωγή σας είπατε ότι το 50% των ατόμων με αναπηρία έχουν πρόβλημα να, να βρουν δουλειά καν. Έχω την εξής ερώτηση τι μέτρα προτίθεστε να υιοθετήσετε ως ε, αρμόδια για την ισότητα σχετικά με την ένταξη και προστασία των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα. Τι εννοώ, μέτρα που να συνάδουν με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τι σχέδια έχετε για να βελτιώσετε την εφαρμογή όλων αυτών στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα ε, ε, βλέπετε νέους τομείς ε, που να καλύπτει η ε, σχετική πρόταση και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς θα συνεργαστείτε με άλλους επιτρόπους για να γίνει προτεραιότητα αυτό το θέμα των ατόμων με αναπηρία. θα καλωσορίσατε την πρόταση να ενταχθεί στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθείας ε, αυτή η ε, αρμόδια υπηρεσία για τα άτομα με αναπηρία, έτσι ώστε να υπάρχει μια γενική επισκόπηση οριζόντια. Απάντηση. Μέχρι το 2020 αναμένεται ε, ένας στους πέντε Ευρωπαίους πολίτες να έχει κάποιο είδους αναπηρία. Όπως είπατε, και η απασχόληση των ατόμων με αναπηρία ε, πάσχει. Είναι πολύ χαμηλή σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει στρατηγική ε, για τα άτομα με αναπηρία 2010-2020, η οποία εκπνέει και πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να αξιολογεί την ε, στρατηγική αυτή. Είναι πολλά τα επιτεύγματα, ε, όπως είναι η πράξη για την προσβασιμότητα που αυτό το καιρό μεταφέρεται, ε, η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η κάρτα αναπηρίας. Τώρα αξιολογούμε τη στρατηγική αυτή και αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι μέλη γενέστε και πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Θα εργαστώ πολύ σκληρά για να σταματήσει η εμπλοκή ε, της οδηγίας για την ίση μεταχείριση και θα εργαστώ για να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Έχουμε τα μέσα λοιπόν και τα εργαλεία για να εργαστούμε σε αυτό το πλαίσιο, το θεσμικό. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η αξιολόγηση των όσων έχουμε καταφέρει με βάση την κείμενη στρατηγική. Συμπληρωματική ερώτηση για ένα λεπτό, Βάρτα. Εσείς στη στρατηγική για το φύλλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμπεριλάβετε και τα άτομα με αναπηρία και στη στρατηγική που προετοιμάζεται εκεί έτσι ώστε να συνάδει με το άρθρο 6 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, όπου καλούνται όλα τα συμβαλόμενα μέρη να ε, αναγνωρίσουν ότι γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία έχουν τετραπλάσιες διακρίσεις Μα τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι οικουμενικά και βασικέ θεμελιώδει ελευθερίε και θα πρέπει όλοι να απολαμβάνουν αυτών των δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Απάντηση. Βεβαίω. Είναι πολύ σημαντική η συμπερίληψη σε όλες τις πολιτικές αυτών των θεμάτων, το mainstreaming όπως λέμε, και θα φροντίσω και τα θέματα αυτά των ατόμων με αναπηρία να αντανακλώνται παντού. Υπάρχει και μια διακομματική ομάδα, ένα intergroup και το φόρουμ το ευρωπαϊκό για άτομα με αναπηρίες. Έχω συνεργαστεί μαζί τους, έχω συναντηθεί μαζί τους. Θέλω φυσικά τα άτομα με αναπηρία να είναι παραστάτες στο πλευρό μου για να μπορέσω να κάνω αυτές τις αλλαγές. Αλλαγές που είναι απαραίτητες για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος. Δεν μπορούμε να αποφασίζουμε για τα άτομα με αναπηρία χωρίς τη δική του συμμετοχή. Και σε οτιδήποτε κάνω, θα συνεργάζομαι μαζί τους. Question one minute. Thank you. Κυρία Γουόλτς, ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Η ισότητα υποτίθεται ότι είναι το θεμέλιο της εξασφάλισης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δίκαιη, όπου οι, προστα... οι αξίες μας προστατεύονται και δεν ισχύουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Όμως θα ξέρετε κι εσείς, θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι πολλή δουλειά πρέπει ακόμα να γίνει για όλα αυτά τα θέματα. Με βάση την προηγούμενη ερώτηση, θέλω να ρωτήσω αν όσοι Επίτροπος για την Ισότητα θα έχετε την ε, ε, αρμοδιότητα για την ισότητα και των ε, ανθρώπων με αναπηρίες και κοινωνικές αναπηρίες. Ένας στους πέντε θα έχει μια αναπηρία μέχρι το 2020. Πώς μπορούμε να βασιστούμε στη νομοθεσία περί πρόσβασης και είστε έτοιμοι να εναρμονίσετε την ε, πρόσβαση ας πούμε στις υπηρεσίες μεταφορών και πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε περισσότερους φοιτητές με αναπηρίες να συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης όπως το Έρασμος. Δύο λεπτά για την απάντησή σας έχετε. Όπως είπα, θα αξιολογούμε την στρατηγική για να δούμε τι έχει γίνει και τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να γίνει καλύτερα ίσως. Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να απεμπλακεί η οδηγία περίσσης μεταχείρισης, γιατί τότε θα έχουμε αποτελέσματα για κάποια από τα ζητήματα που αναφέρατε, αλλά... Και επίσης η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία είναι η βάση για την εργασία που θα κάνουμε και όπως είπα και προηγουμένως θέλω να συνεργαστώ με όλους όσους εκπροσωπούν ε, ενώσεις αναπήρων. Το έχω κάνει άλλωστε και παλιότερα. Είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας πολιτικής. Και όπως είπατε, δικαίως πολλά πρέπει ακόμα να γίνουν και προσβλέπω και στο θέμα του mainstreaming για τα θέματα της αναπηρίας σε όλες τις ε, πολιτικές της Επιτροπής, χρησιμοποιώντας δηλαδή τις ε, ε, ομάδες, τις ειδικέ που υπάρχουν, ώστε μαζί με το mainstreaming για την ισότητα να έχουμε και mainstreaming για τις ανθρώπους με αναπηρίες. Μάλιστα, επερώτηση. Ξέρω πως στηρίζεται την απόφαση της Προέδρου Βαντελάινα να δώσει το χαρτοφυλάκιο που προστατεύει την ευρωπαϊκή, ε, τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, ε, ε, να φτιάξει μάλλον χαρτοφυλάκιο για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και το υποστηρίζω. Αλλά ξέρω πως υπάρχει πολλή, πολλή συζήτηση για όλα αυτά. Όμως εσείς τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση του θέματος των αδικημάτων, των εγκλημάτων μίσους επιγραμμικά και ε, στην πραγματική ζωή. Κοιτάξτε, ο, ο λόγος μίσους για τον οποίο μιλάτε είναι βεβαίως κάτι πολύ πολύ σοβαρό και μάλιστα καθώς κρατάει πολύ κόσμο μακριά από την τεχνολογία. Για παράδειγμα, κάποιες γυναίκες ε, δεν χρησιμοποιούν ε, τεχνολογία λόγω του μίσους ή ανθρώπων ή πραγμάτων που τα οποία έχουν υποφέρει. Ε, ε επίσης, Κάποιες φορές ε, βλέπουμε πως οι γυναίκες ε, στην τεχνητή νοημοσύνη ή στην ε, τεχνολογία της πληροφορίας είναι λιγότερες γιατί γι' αυτό το λόγο. Εγώ θα συνεργαστώ με τους επιτρόπους που είναι αρμόδιοι για αυτό το τομέα. Η κυρία Πιτσέρνο. Ένα λεπτό έχετε για την ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητή Επίτροπε, εσείς παραθέσατε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 ε, κύρωση της σύμβασης της ε, Κωνσταντινούπολης ως προτεραιότητα για την Κομισιόν. Φυσικά χαιρόμαστε για αυτή σας ε, την δήλωση γιατί πιστεύουμε πως η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι ένα σημαντικό μέτρο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Γνωρίζουμε όμως ωστόσο πως και η διαδικασία συνυπογραφής έχει προλοκαριστεί λόγω κάποιων συντηρητικών κυβερνήσεων που εδώ και χρόνια εμποδίζουν και καθυστερούν την κύρωση ιδεολογικούς λόγους. Θα ήθελα να γνωρίζω πώς πιστεύετε ότι θα ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και θα θέλαμε να ξέρουμε αν πιστεύετε πως είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή ώστε να προταθεί οδηγία της Ένωσης που θα αντιμετωπίζει τη βία κατά των γυναικών με συνεπή και συνολικό τρόπο σε όλα τα κρατημέλη. Εσείς στις ε, γραπτές σας απαντήσεις αναφερθήκατε στην πρόθεσή σας να αντιμετωπίσετε και τους νέες αναδυόμενες μορφές ε, έμφυλης βίας, ειδικά αυτές που γίνονται επιγραμμικά. Ποιος θα είναι ο τρόπος και ποιες θα είναι, ποια θα είναι τα μέτρα για να αντιμετωπίσετε αυτή την πραγματική ε, πληγή κατά των γυναικών. Πιστεύετε πως ε, μια τέτοια οδηγία θα πρέπει να περιλαμβάνει και αυτού του είδους της μορφές βίας. Μάλιστα, απάντηση δύο λεπτά. Ξέρουμε ότι η κατάσταση σήμερα είναι ότι μία στις τρεις γυναίκες θα υποστούν βία λόγω και μία στις τέσσερις ε, οικιακή βία, οικογενειακή βία και το κόστος ε, αυτών των ε, επεισοδίων είναι 226 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ε, συνδυάζει διαφόρους τομείς εθνικών και ενωσιακών αρμοδιοτήτων. 20 κράτη, 21 μάλιστα, κράτη-μέλη, την έχουν επικυρώσει. Αλλά θα γνωρίζετε επίσης ότι κατά την ε, Προεδρία της χώρας μας εργαστήκαμε για να υπάρξουν περαιτέρω υπογραφές και η Ένωση υπέγραψε αυτή την σύμβαση. Όλοι θέλουμε να υπάρχει και πρόληψη και προστασία των θυμάτων και διώξεις ε, των υπευθύνων και ολοκληρωμένες πολιτικές. Θα ε, συζητήσω με τα απρόθυμα κράτη-μέλη, θα επισκεφθώ αν χρειαστεί και τις πρωτεύουσε για να επιδιώξω να υπάρξει συμφωνία για τη σύμβαση αυτή. Για μένα είναι πολύ σημαντική. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχουν αντιστάσεις. Υπάρχουν ίσως διαφορετικές απόψεις για κάποιες διατυπώσεις αλλά άμα δει κανεί ε, τις στατιστικές, μία στι τρεις γυναίκε έχουν υποστεί βία λόγω φύλου. Πώς είναι δυνατόν να μην δεσμευτεί κανεί να κάνει περισσότερα, να επικυρώσει η Ένωση δηλαδή αυτήν την σύμβαση. Συμπληρωματική ερώτηση ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ επανέρχομαι στο θέμα τη οδηγία, που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει συνολικά το θέμα τη βία κατά των γυναικών. Εσεί αναφέρατε σημαντικά ε, στοιχεία ότι κάθε γυναίκα, είτε είναι πλούσια, είτε είναι φτωχή, είτε είναι ισχυρή, διάσημη ή άγνωστη, κάθε γυναίκα, σε όποια και είναι η θρησκεία της, και η θρησκεία της, η πίστη της κτλ. Καθημερινά, κυρία υποψήφια επίτροπη, ε, υπόκειται σε διάφορες μορφές βίας. Είτε είναι σωματική, είτε είναι ε, ε, ρητορική, είτε είναι οτιδήποτε. Είναι κάτι το απαράδεκτο για την ελευθερία μας και για τη ζωή μας. Γι' αυτό σας ζητώ να δράσετε με συγκεκριμένο τρόπο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απόλυτα. Αλλά... Ε, μα, ε, gender equality strategy Στην στρατηγική για την ισότητα των φύλων θα υπάρχει και δηλαδή θα αντιμετωπιστεί μάλλον και το θέμα της βίας. Ε, τώρα, εγώ θέλω να πετύχω, θέλω να πετύχω στο να καταφέρω να ε, κυρωθεί η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα υπάρχει και η οδηγία και τα δικαιώματα των θυμάτων που μπορεί να ενισχυθεί. Υπάρχει επίσης ε, Μπορούμε επίσης να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε αδίκημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο την βία κατά των γυναικών, αλλά δεν θέλω να στραφώ προς τα εκεί. Θέλω πρώτα να προσπαθήσω να εξασφαλίσω την κύρωση της σύμβασης. Ευχαριστώ. Η κυρία Λάγκεντζιπ, παρακαλώ, ένα λεπτό για την ερώτησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ως πράσινοι και εγώ ως η πρώτη γυναίκα που έχω ορατή αναπηρία, χαιρετίζω το γεγονός ότι η ισότητα και η συμπερίληψη είναι προτεραιότητα της Κομισιόν. Θα πρέπει σε όλες τις πολιτικές μας να ε, υπάρχει αυτή η διάσταση. Χαίρομαι που εσείς κυρία Αντάλη ιδιαίτερα λέτε ότι είναι οριζόντια αρμοδιότητα και θέλετε να εφαρμοστεί πλήρως η Σύμβαση των Ηνωμένων για τα άτομα με αναπηρία. Όλα αυτά είναι βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω παρακαλώ να μου απαντήσετε με ναι ή όχι στην απλή ερώτηση. δεν διατεθειμένοι να θέσετε βέτο σε οποιαδήποτε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν συμπεριλαμβάνει αυτά τα δικαιώματα. Όλες τις νομοθετικές προτάσεις και όλες τις προτάσεις για χρηματοδότηση θα τις σταματάτε αν δεν περιλαμβάνουν αυτή τη διάσταση. Θα ελέγξετε όλες τις προτάσεις της Κομισιόν για να δείτε εάν εφαρμόζουν αυτήν τη Σύμβαση των Εθνών. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά για την απάντησή σας παρακαλώ. Η απάντησή μου είναι ναι. Ναι, δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι είναι στις δυνατότητές μου, ούτως ώστε να εφαρμοστεί αυτή η σύμβαση πλήρως και χωρίς εξαιρέσεις. Επίσης, θα κάνω ό,τι μπορώ, ούτως ώστε τα θέματα αναπηριών να είναι σε όλες τις πολιτικές. Μέσω αυτής της ειδική ομάδας, Task Force, και θέλω να επεκταθεί η αρχή του ελέγχου για θέματα ισότητας. Και θα συνεργαστώ πολύ στενά με τη διαπολιτική ομάδα για τις ε, αναπηρίες και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις ε, αναπηρίες. Παρακαλώ, συμπληρωματική ερώτηση, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντάλη. Είπατε ότι πρέπει να προσέξουμε ότι πρέπει να συμμετέχουν στα διάφορα εγχειρήματα τα άτομα με αναπηρία. Αυτό είναι πολύ σωστό. Αυτό ανταποκρίνεται στο αίτημα των ατόμων με αναπηρία τίποτα για μας χωρίς εμάς. Πρέπει να συμμετέχουν λοιπόν τα άτομα με αναπηρία για κάθε απόφαση που τα αφορά εμείς ως πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα τα παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά αυτά και τη σημερινή σας δέσμευση θα στις υπενθυμίζουμε. Πρέπει να είστε θέματο, ε, θεματοφύλακα των θεμάτων αυτών για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό απάντηση. Μα φυσικά θα με παρατηρείτε. Θα με συμβουλεύετε επίσης. Όπως είπα, θέλω συνεχή διάλογο με το Κοινοβούλιο. Θέλω πραγματικά να συνεργαστώ ενεργά με όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου για τα διάφορα θέματα. Είναι πολύ σημαντικό τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με την κοινωνία των πολιτών να συμμετέχουν, να ακούμε οι μεν τους δε, να ανταλλάσσουμε ιδέες, να επικρίνουμε οι μεν τους δε. Είναι πολύ σημαντικό να μας επικρίνεται. Η επικοδομητική κριτική οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπρούνα. Κυρία Νταλή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θελήσαμε να ενισχύσουμε τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας. Να βρούμε έναν τρόπο για να ενισχύσουμε τα θύματα, ιδιαίτερα της ενδοοικογενειακής βίας, να ενισχύσουμε την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων. Πλην όμως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά τη συζυγική βία, αυτό το θέμα δεν έχει συζητηθεί ε, τουλάχιστον επαρκώς, ιδιαίτερα ε, τι γίνεται με τα παιδιά που είναι θύματα όταν η μητέρα τους υφίσταται τη βία. Μιλήσατε για το λόμπι, ΛΟΑΤΚΙ, το οποίο ενισχύεται, ενώ τα παιδιά που είναι θύματα αυτής της ενδοκιογενειακής βίας δεν έχουν καμιά επιτροπή να τα υποστηρίζει ούτε στο Κοινοβούλιο ούτε στην Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να είναι ε, το συμφέρον τους ε, ύψιστο και το ενδιαφέρον μας επίσης. Εσείς που φιλοδοξείτε να γίνετε επίτροπος ισότητας, ε, τι σκοπεύετε να κάνετε για να καλύψετε αυτό το έλλειμμα και αυτά τα παιδιά που είναι ξεχασμένα. Απάντηση. Όταν συζητούμε για οικογένειες, για ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Όταν μιλούμε για οικογένειες ε, προβληματικές, ε, δυσλειτουργικές, με προβλήματα βίας στο εσωτερικό τους, προφανώς και σκεφτόμαστε και τα παιδιά. Θύματα είναι τα παιδιά τέτοιων καταστάσεων. μέσα στις οποίες ζουν. Και γι' αυτό θα πρέπει να απολαμβάνουν προστασίες και να ε, απομακρύνονται από το δράστη αυτών των κρούσματων βίας. Μαζί με το θύμα, το φυσικό θύμα που είναι συνήθως η μητέρα τους, αλλά και τα παιδιά θα πρέπει να προστατεύονται από εκείνον που βιοπραγεί εις βάρος τους. Εγώ θα συνεργαστώ με την Επίτροπο που είναι αρμόδια ε, για τα παιδιά ε, και θα συνδυάσουμε έτσι, την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, της ενδοοικογενειακής βίας ε, με τα δικά της θέματα για την προστασία των ανηλίκων και τα δικαιώματα των παιδιών. Φυσικά, είναι απόλυτη ανάγκη η προστασία των παιδιών σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί είναι τα πιο ανυπεράσπιστα μέρη αυτής της ε, εξίσωσης. Σας ευχαριστώ που το θέσατε. Και στη στρατηγική μας, εκεί που ε, κάνουμε λόγο για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, συμπεριλαμβάνουμε και τα παιδιά. Συμπληρωματική ερώτηση για ένα λεπτό, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας γιατί προφανώς ε, αυτή η υπόθεση ε, έχει τη θέση της σε συζήτηση αυτή αδιαφεσβήτητα και σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας που δηλώνετε ότι θα δείξετε στο μέλλον σε αυτό το πρόβλημα. answer or we get... Να απαντήσουμε ή να προχωρήσουμε. Κυρία Ραφάλσκα, παρακαλώ ένα λεπτό. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, σας έχουν εμπιστευτεί το καθήκον αντιμετώπισης κάθε είδους ε, ανισότητας και διακρίσεων. Η Ένωση βασίζεται σε χριστιανικές αρχές. Αλλά τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε αύξηση των διακρίσεων, ακόμη και απολύσεις επειδή κάποια άτομα φοράνε χριστιανικά σύμβολα ή ενστερνίζονται χριστιανικές αρχές και υπάρχουν και επιθέσεις κατά χριστιανών ή μάλλον ε, υπάρχουν κατηγορίες κατά χριστιανών από ορισμένου που λένε πως είναι κατά των διακρίσεων. οι οποίοι κάνουν διακρίσεις στην ουσία κατά των χριστιανών. Πώς θα προστατεύσετε λοιπόν τα δικαιώματα των χριστιανών κατά των διακρίσεων. Παρακαλώ. Κυρία Υποψηφία Επίτροπε. Θα εργαστώ για την οδηγία κατά των διακρίσεων η οποία αναφέρεται για διακρίσεις, ε, για λόγους ηλικίας, πεπιθήσεων, θρησκείας, ε, αναπηριών και σεξουαλικού προσανατολισμού. Θα περιμένω να γίνει το Συμβούλιο για την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική, την υγεία και, ε, και τα θέματα καταναλωτών που θα γίνει τον Οκτώβριο για να δω τι θα γίνει με αυτή την οδηγία η οποία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είναι μπλοκαρισμένη. Αν ε, καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο για αυτή την οδηγία, θα βελτιώσουμε την κατάσταση. Θα βοηθήσουμε όλα αυτά τα θύματα διακρίσεων και για το λόγο που αναφέρατε. Προφανώς, είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχουν και φορείς κύρους στα κράτη-μέλη που να ασχολούνται με τα θέματα αυτά. για να αντιμετωπίσουν ακριβώς τα διάφορα θέματα που προκύπτουν στην κοινωνία μας. Και διάφορες χάρτες ισότητας είναι σημαντικό να υπάρχουν. Αλλά το πιο σημαντικό από την πλευρά μου αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσει αυτή η οδηγία κάτω των διακρίσεων. Με πολύ ενθουσιασμό περιμένω να γίνει αυτό το Συμβούλιο αργότερα το μήνα αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Ραφάλσκα, σημαντική ερώτηση, ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, γνωρίζετε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου για τις Βρετανικές αερογραμμές για διακρίσεις κατά των εργαζομένων στις Βρετανικές αερογραμμές για λόγους ε, θρησκείας. Στην Πολωνία έχουμε μια υπόθεση όπου ένας εργαζόμενος του IKEA υπέστη κυρώσεις επειδή έκανε παράθεση από τη βίβλο. Δεν θεωρείτε ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Δεν καταλαβαίνετε τι διακυβεύεται. δεν είναι θέμα μόνο των χριστιανών. Είναι προστασία γενικά δημοσίων ελευθεριών. Κοιτάξτε. Ως εμείς είσαι μη ποιήσεις. Αυτή είναι η αρχή μου. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η οδηγία κατά των διακρίσεων είναι σημαντική. Είναι θέμα ε, ίση αντιμετώπιση όλων ανεξάρτητα από τις πεπιθήσεις, τη θρησκεία, την ηλικία, το σεξουαλικό προσανατολισμό. Α εργαστούμε λοιπόν για να προχωρήσει αυτή η οδηγία. Τώρα η κυρία Βόζομπερ Βριονίδη. Παρακαλώ. Πέρα σας ως, είμαι Ελληνίδα δικηγόρος επί τρεις δεκαετίες και αισθάνομαι την υποχρέωση να σας πω ότι θεωρείται πλήγμα για τη δημοκρατία στη χώρα σας και για το κράτος δικαίου το γεγονός ότι είναι ακόμη ανεξιχνίαστη η στιγερή δολοφονία της Δάφνης Καλιτσία, όχι γιατί ήταν γυναίκα, αλλά γιατί ήταν μια αγωνίστρια της αλήθειας και υπηρετούσε την αποκαλυπτική δημοσιογραφία. Ως προς την ερώτησή μου, παρακαλώ, θέλω να σας μιλήσω για τη γυάλινη οροφή είχα την ευθύνη να έχω την έκθεση στην περασμένη περίοδο και ξέρετε πολύ καλά ότι αναφέρεται στις ανισότητες που ορθώνονται στις γυναίκες καριέρας, στην επιστήμη και στην ε, τεχνολογία, στην έρευνα, όπου υπάρχει και μια αύξηση συμμετοχής γυναικών. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσον έχετε μια εμβληματική πρωτοβουλία ή με διαφορετικό τρόπο χρήση των ήδη υπαρχουσών πολιτικών, ώστε να αντιμετωπιστεί η εξάλληψη των προκαταλήψεων αντιλήψεων και των στερεοτύπων που εμποδίζουν την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά. Σας ευχαριστώ. Answer two minutes. Η απάντηση δύο λεπτά παρακαλώ. Είχα την ευκαιρία να πω προηγουμένως ότι οι έρευνες για τη γυναικοκτονία εις βάρος της Δάφνης Καρό Αναγκαλίσια συνεχίζονται. Συνελήφθησαν ε, και απεγγέλθηκε κατηγορία σε τρία άτομα ήδη από τις πρώτες μέρες. Σε ό,τι αφορά τη γυάλινη οροφή, πραγματικά υπάρχει ακόμα και ε, πραγματικά πολύ ήπια ε, το λέμε Είμαι ακράδαντα πεπισμένη ότι θα πρέπει να εξαλείψουμε τα στερεότυπα και να συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες ε, σε αυτές τις θέσεις. Την χάνει εγώ προσωπικά να ε, προώθησα τη Διεθνή ημέρα για τα κορίτσια και τις γυναίκες στις επιστήμες στα Ηνωμένα Έθνη. 11 Φεβρουαρίου είναι η μέρα ε, όπου εορτάζουν τα Ηνωμένα Έθνη, ε, μια δική μου πρόταση. Καταλαβαίνετε πόσο με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι θετικές επιστήμες και πόσο θέλω να ε, συμμετέχουν, να κορίτσια να σπουδάζουν θετικές επιστήμες και οι γυναίκες που ήδη είναι στις επιστήμες αυτές να έχουν ηγετικές θέσεις και για τα παιδιά και να δημιουργούνται νέα μοντέλα. Βεβαίως έχουμε αυτά τα στερεότυπα που θα πρέπει να καταπολεμήσουμε. Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Να πατάξουμε στη στρατηγική για το φύλλο. Αυτό έψαχνα και δεν μου ερχόταν η έκφραση. Στρατηγική για το φύλλο. Follow-up question. Ρωματική ερώτηση παρακαλώ για την απάντηση. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά ε, πάλι στο θέμα της ισότητας, εφόσον πρόκειται να είστε ε, επίτροπος στην ισότητα, για το θέμα του χάσματος που υπάρχει στην συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή εποχή. Το χάσμα αυτό θέλει μια ειδική αντιμετώπιση και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε κάποια εμβληματική πρωτοβουλία σε αυτό, ούτω ώστε να μπορούμε την επόμενη μέρα να πούμε ότι υπάρχει μια ισότιμη εκπροσώπηση στο, στους τομείς της τεχνολογίας, των πληροφοριών πληροφοριών, των επικοινωνιών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διότι είναι δεδομένο ότι σε αυτό το τομέα υπάρχουν και υψηλέ αμοιβέ και η εκπροσώπηση των γυναικών είναι στα κατώτατα επίπεδα, κάτι που δεν τιμά τη δημοκρατία μας και το κράτος δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Yes, uh, uh, Μάλιστα. Η πληροφορική ε, δεν μπορεί να παραμείνει ε, τσιφλίκι ανδρικό. Και είναι και πολύ καλοπληρωμένες οι θέσεις αυτές, όπως πολύ καλά είπατε, και τα επαγγέλματα. Και αυτό συνεχίζει να έχει επιρροή ε, στο μισολογικό χάσμα και την ψαλίδα αυτή. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Θα πρέπει όμως οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα στερεότυπα. Οι γυναίκες γιατί δεν κατευθύνονται, δεν καθοδηγούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό σας ανέφερα ε, τη Διεθνή ημέρα κοριτσιών και γυναικών στις θετικές επιστήμες. Και σε ό,τι αφορά και την ε, πανεπιστημιακή ακαδημιακή πορεία, ξέρω περίπτωση όπου όταν δεν ήταν υποχρεωτικά τα μαθήματα αυτά των ε, επιστημόνιων, ε, ε, τα κορίτσια δεν τα επέλεγαν. Όταν ήταν υποχρεωτικά, τα κορίτσια ήταν καλύτερες μαθήτριες σε αυτά τα μαθήματα. Άρα ε, το θέμα είναι τα στερεότυπα και αυτός ο επαγγελματικός προσανατολισμός που δεν οδηγούν τα κορίτσια προς τις κατευθύνσεις αυτές. That's why we have the digital gap also in... οπότε πραγματικά και εκεί υπάρχει ένα χάσμα. Η κυρία Ροντρίγκε, παρακαλώ, ένα λεπτό για την ερώτησή σας. Ε, gracias, Ελέκτα. Ευχαριστώ, κυρία υποψήφια επίτροπε και καλή επιτυχία στην ε, υπεράσπιση της ισότητας. Το θέμα των ε, του μίσου κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜΑ, παίρνει διάφορες μορφές ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, προφορικές προσβολές, ε, έλλειψη επίσης ε, πρόσβαση σε πολλές από τις παροχές. Έγινε λόγος για μια οδηγία για την κατάργηση των διακρίσεων. Φαντάζομαι ότι και ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι ένας από, τους, από τους λόγους για τους οποίους τον μπλοκάρισαν τα κράτη-μέλη. Ποια είναι η στρατηγική σας για να ξεπεράσετε τον μπλοκάρισμα και ποια είναι η στρατηγική σας για να δουλέψετε με τα κράτη-μέλη ώστε να επιτύχετε να υιοθετήσουν ε, τα αίτια ε, ταυτότητας φύλου ε, στη ε, στάση τους. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά για την απάντησή σας. Εγώ να σας εξηγήσω ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι επιλογή. Αν αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο μπλοκάρει η οδηγία, θα ήθελα αυτό να το καταλάβω καλύτερα, γιατί δεν το καταλαβαίνω αν όντω αυτό είναι ο λόγος. Αλλά υπάρχουν περισσότερα προβλήματα. Σε κάποια κράτη-μέλη, λιγότερο από το 50% των ανθρώπων πιστεύουν πως οι ε, ΛΟΑΔΜΑ θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους ετεροφιλόφιλους. Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο μέσα εργαζόμαστε. Όπως ξέρετε, υπάρχει ε, ο κατάλογος δράσεων που αφορά τη βελτίωση των δικαιωμάτων των ανθρώπων ε, ΛΟΑΔΜ και των οικογενειών τους, παρακολούθηση της ε, εφαρμογής, της επιβολής μάλλον των ισχυουσών οδηγιών και δικαιωμάτων. Πολλά γίνονται δηλαδή. Τώρα θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των ε, δράσεων και μετά στη συνέχεια να προτείνουμε και ισχυρά μέτρα. Αλλά όπως είπατε πρέπει να προχωρήσουμε αυτή την οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων. Αυτό είναι ο τρόπος που θέλω εγώ να προχωρήσω και που θέλω να προσπαθήσω να κατανοήσω γιατί είναι τόσο δύσκολο να ξεμπλοκαριστεί αυτή η κατάσταση. Επίσης να αναφέρω την ομάδα υψηλού επίπεδου για την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Ε, ε, η υπερώτηση τώρα, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να αγωνιστούμε για τους πιο ευάλωτους και για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είπατε στην εισήγησή σας. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η δική σας νόμη για την πρωτοβουλία που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση Spot με 50 εκατομμύρια ευρώ για να ξεκινήσει και να βοηθήσει ένα παγκόσμιο κίνημα κατά της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγγυηθούμε την υπεράσπιση των γυναικείων δικαιωμάτων έναντι της θεσμικής, ατομικής και διαθρωτικής βίας, ανεξάρτητα από την νομική της κατάσταση, δηλαδή το καθεστώς, είτε είναι δηλαδή γυναίκες ε, πρόσφυγες ή άνευ ε, χαρτιών. Απάντηση. Όπως γνωρίζετε, Είμαστε δεσμευμένοι για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και έχουμε μέσα ε, τα οποία, με τα οποία θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικές πραγματικότητες. Ε, ε, θα πρέπει να δουλέψουμε εσωτερικά και εξωτερικά και να στηρίξουμε πρωτοβουλίες νομοθετικές και μη όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των ε, διαφόρων ε, ανθρώπων και φυσικά θα εργαστούμε στους τομείς που εσείς αναφέρατε και θα πιέσουμε ώστε να προχωρήσουν και να προωθηθούν τα δικαιώματα των διαφόρων ομάδων ανθρώπων για τις οποίες μιλήσατε. Κύριος Νικολάου, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα ελληνικά, προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσει προωθούν την πολιτική τη συμφιλίωση επαγγελματική και οικογενειακή ζωή για να διαχειριστούν τι συνέπειε από την αύξηση τη γυναική απασχόληση και την έλλειψη μέτρων στήριξη τη οικογένεια. Κομβική θέση σε αυτέ τι συγκεκριμένε κατευθύνσει κατέχει η πλήρη ευελιξία χρόνου και χώρου εργασία που σπάει κάθε κανονικότητα στα ωράρια, οδηγεί στον κατακαιρματισμό τη κοινωνική ζωή τη εργαζόμενη γυναίκα μητέρα το ενδιαφέρον για την προστασία τη μητρότητα φτάνει μέχρι το σημείο που τα όποια μέτρα δεν αποτελούν κόστο για τι μεγάλε επιχειρήσει. Στο έδαφο τη πλήρου ευελιξία των εργασιακών σχέσεων, 71% των εργατοϊπαλλήλων γυναικών στερούνται ακόμα και τι πενιχρέ άδειε και επιδόματα μητρότητα, τα οποία απαιτούν ορισμένο αριθμό ημερομισθείων. Μεγάλο μέρο των εγγύων στερούνται τη στοιχειώδη προστασία από απόλυση, όπω υπογραμμίζουν επίσημα στοιχεία του ILO. Πώ τοποθετήστε στην κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασία, για την νομοθετική κατοχήρωση τη κοινωνική προστασία τη μητρότητα για όλε τι μισθωτέ, ανεξαρτήτω σχέση εργασία, για την απαγόρευση απόλυση εγγύων. Ευχαριστώ. The answer, two minutes. Παρακαλώ δύο για την απάντηση. Η προστασία των συνθηκών ε, απασχόλησης και των εργαζομένων Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Όπως είπατε. Είναι θέμα συνδυασμού ε, προσωπικής, ιδιωτικής δηλαδή και πραγματικής ζωής για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των οικογενειών. Αλλά ακόμη υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. τα θέματα που αναφέρατε. Είναι θέματα που θα συζητήσω με τον ε, υποψήφιο επίτροπο Σμιτ. Θέλουμε να δούμε τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση για τις συνθήκες εργασίας. Για να δούμε τι θα μπορούσαμε να προτείνουμε για να εντοπίσουμε τα θέματα που αναφέρατε. Κύριε Νικολά, συμπληρωματική ερώτηση, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για να κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα τα ζητήματα. Πώς τοποθετήστε στο ότι με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που γνωστοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου του 2018 που επιτρέπει την απόλυση εγγύων εργαζομένων στο πλαίσιο των ομαδικών απολύσεων ανοίγει στην πραγματικότητα ο δρόμος για περαιτέρω εξαιρέσεις που θα οδηγήσουν στο να μην υπάρχει καμία μα καμία προστασία των εγγύων και των νέων μητερών στον, στην εργασία τους. The answer, one minute. Ένα λεπτό για την απάντηση, παρακαλώ. Θα πρέπει να δω την απόφαση αυτή του δικαστηρίου και με χαρά να συναντηθούμε και να το συζητήσουμε. Αλλά φυσικά οι έγκυες θα πρέπει να έχουν προστασία. Η κυρία Σαλίμπα, ένα λεπτό για την ερώτησή της. Ο κύριος Σαλίμπα. Και είμαι Μαλτέζος και είμαι πολύ περήφανος που έχετε επιλεγεί για το χαρτοφυλάκιο της ισότητας. Κατά τη σταδιοδρομή σας στη Μάλτα ήσασταν υπεύθυνοι για αυτά τα θέματα ακριβώς και καταφέρατε να επιτύχετε μια κοινωνική επανάσταση. Καταφέρατε δηλαδή η χώρα μας να γίνει υπόδειγμα για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την προστασία των μειονοτήτων. Ελπίζω λοιπόν ότι στην επόμενη πενταετία θα καταφέρετε να προωθήσετε την ισότητα στην Ευρώπη. Η οδηγία για το συνδυασμό ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου έχει εγκριθεί και η σοσιαλιστική ομάδα ήταν πρωτοπόρα στη στήριξη αυτής τη οδηγίας. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου πολλά κράτη-μέλη τώρα παρεμποδίζουν την εφαρμογή της. Συμφωνώ ότι ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμοστεί τάχιστα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι πρέπει να ε, διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του για να συμπεριλάβει και τα δικαιώματα των ε, ελευθέρων επαγγελματιών και των γονέων που υιοθετούν παιδιά. Απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ναι, προφανώς, όπως ήδη είπα, απαντώντας τον κύριο Κάζα, θα συνεργαστώ για να εφαρμοστεί σωστά αυτή η οδηγία. Τώρα για την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή τη. Εγώ θεωρώ ότι τώρα πρέπει να εστιάσουμε κυρίως ε, στην εφαρμογή για τα επόμενα τρία χρόνια. Να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι η οδηγία όπως έχει θα εφαρμοθεί πλήρως και σωστά από τα κράτη-μέλη. Και μετά, επειδή ούτω ή άλλω υπάρχει ρήτρα αναθεώρηση τη οδηγίες, μετά λοιπόν, εάν χρειάζεται, θα αξιοποιήσουμε αυτή τη ρήτρα για να δούμε εάν και κατά πόσο πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής της. Για να συμπεριλάβουμε και τα δικαιώματα που αναφέρατε. Αλλά για τα επόμενα τρία χρόνια το βασικό είναι να εφαρμοστεί σωστά σε κάθε κράτος μέλος η οδηγία αυτή. Συμπληρωματική ερώτηση, ένα λεπτό. Ναι. Ένα άλλο θέμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Τα άτομα με αναπηρίες. Η στρατηγική μας για τη δεκαετία 10 και 20 ήταν να εφαρμόσουμε την Σύμβαση των Ηνωμένων για τα άτομα με αναπηρίες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Πώς θα διασφαλίσετε να συμπεριλαμβάνετε σε όλους τους τομείς πολιτικής το θέμα αυτό. Θα φροντίσετε να υπάρξει αναθεώρηση της εφαρμογή για να διασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή αυτής της ε, σύμβασης. Και θα θέλατε να έχει πιο φιλόδοξου στόχου για τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα δέκα χρόνια αυτή η σύμβαση. Σε ευχαριστώ για την προσωπική σα δέσμευση και δουλειά, ούτω ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι ενώσει των ατόμων με αναπηρία στι συζητήσει για τα θέματά του. απάντηση. Σας ευχαριστώ. Τώρα ε, πλησιάζουμε το τέλος της περίοδου εφαρμογή αυτής της, ε, της πρώτης περίοδου εφαρμογή αυτής της σύμβασης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε περαιτέρω. Να κάνουμε μια αξιολόγηση για το πώς λειτουργήσε την ε, τρέχουσα δεκαετία η εφαρμογή της σύμβασης. Στην αξιολόγηση θα δούμε σαφέστερα την κατάσταση θα δούμε ποιες ήταν οι αδυναμίες ε, που μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις. Και τώρα για τη συμπερίληψη του θέματος αυτού σε όλα τα θέματα, σε όλους τους ε, κλάδους πολιτικής. Θα διασφαλίσουμε ότι θα γίνει αυτό. Θα το θέσουμε σε όλες τις γενικές διευθύνσεις, θα διασφαλίσουμε ότι θα το λαμβάνουν υπόψη όταν διατυπώνουν προτάσεις. Ούτως ώστε αυτή η σύμβαση να είναι τμήμα όλων των πολιτικών, στο επίκεντρο. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ειδική ομάδα και όλα αυτά που αναφέρατε θα φροντίσουμε να είναι καθημερινό μέλημά μας στην εργασία της Επιτροπής. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά για τα θέματα ισότητα. Η κυρία Σταρά Φεραγκότ, ένα λεπτό για την ερώτησή σα. Να ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, κυρία Υποψήφια Επίτροπε, ευχαριστώ. Σύντομα δύο ερωτήσει. Πρώτον, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Φύλλο. Δεν λαμβάνει υπόψη τη την ανάπηρη γυναίκα. Κανονικά θα πρέπει να αυξηθεί η μητρική άδεια για τη γυναίκα με αναπηρία. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Αναπηρίες ούτε αυτή λαμβάνει υπόψη την ανάπηρη γυναίκα. Άρα θα πρέπει να κάνουμε μια στρατηγική καινούργια και να μην ε, καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Νέα στρατηγική αξιολόγηση και ξανά νέα στρατηγική, τέλειωσε η θητεία. Θα πρέπει να δούμε τι έχει κάνει η ε, Ευρωπαϊκή Πράξη για την προσβασιμότητα. Ε, τρία χρόνια για να μεταφερθεί και άλλα τρία για να εφαρμοστεί και μάλιστα ορισμένες υπηρεσίες ε, καθυστερούν μέχρι το 2030. Και εδώ έχουμε τώρα και την κλιματική αλλαγή. Ας τα αλλάξουμε. Ε, θα πρέπει να αλλάξουμε τις συνειδήσεις με τους νόμους. Δύο λεπτά για την απάντηση. Μάλιστα. Το θέμα της αναπηρίας θα ενταχθεί στη στρατηγική του φίλου. γιατί ακριβώς αυτό είναι η ένταξη ε, της αναπηρίας σε όλα τα πεδία της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά για τη στρατηγική αυτή καθ' αυτή θα πρέπει πρώτα να την αξιολογήσουμε. Δεν λέω ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2030. Αυτό που λέγω είναι ότι πριν δεσμευτούμε να φέρουμε κάτι άλλο, πρέπει πρώτα να αξιολογήσουμε αυτό που έχουμε, αυτό που είχαμε και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, αντλώντας τα διδάγματα της εφαρμογής της προηγούμενης στρατηγικής. Question, one minute. Ε, ερώτηση, ένα λεπτό. Η πράξη για ε, την προσβασιμότητα έχει αφήσει απ' έξω διάφορες υπηρεσίες στέγασης, εστίασης, ε, ε, τοπικές συγκοινωνίες, ένα σωρό άλλα πράγματα, τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στα θέματα ισότητας, ας μην δημαγωγούμε, γιατί μπορεί να είναι καλές συζητήσεις και ξαφνικά μέσα στα θέματα μπλέκεται η άμβλωση και τα μπερδεύει όλα και διαπληκτιζόμαστε. Ας αφήσουμε τις ιδεολογίες και να ασχοληθούμε με αυτά που μας ενώνουν, γιατί, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα που δεν έχουν ιδεολογία, ούτε αυτά ούτε η ειρήνη. Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο Θα πρέπει να τα αναλύσουμε όλα αυτά και να τα αξιολογήσουμε. Και για όλους αυτούς τους λόγους που εσείς αναφέρατε, για να δούμε πώς ε, μπορούμε να συνεχίσουμε από όλα αυτά που αναφέρατε, που είναι πάρα πολύ εύστοχα όλα, και τα έχω ακούσει κι εγώ όταν συναντήθηκα ε, με ε, τους εκπροσώπους στο ΜΚΟ, ακριβώς τα ίδια λέτε κι εσείς. Όσα μου είπαν εκείνη, τα έχω υπόψη μου. Και κατά τη διάρκεια αυτής της αξιολόγησης ακριβώς θα τα λάβω υπόψη όλα αυτά που λέτε, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά και εύστοχα. Ευχαριστώ. Madame Rodriguez Palop. Your... Η κυρία Ροντρίγκεθ Παλόπ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές οικιακά εργαζόμενες ε, διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να είναι αντικείμενο εκμετάλλευση και δεν ε, προστατεύονται από κανόνες απασχόλησης. Πολλές φορές ε, τις κακομεταχειρίζονται τα αφεντικά τους και κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους πολύ εύκολα και αυτό μπορεί να σημαίνει ιδίω για τις μετανάστριες και την απέλαση. Πρέπει να εργάζονται γιατί δεν έχουν καμία προστασία μέχρι 18 ώρες την ημέρα με πολύ ξεκούραση και δεν έχουν σχεδόν καθόλου μέρες ξεκούρασης. Θα λάβετε μέτρα για να βελτιώσετε τις ηθίκες εργασίας αυτών των εργαζομένων. Θα προωθήσετε την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη και ναι, πριν, μετά την έγκριση από το Συμβούλιο τη σύμβαση του Διεθνού Οργανισμού Εργασία για τι οικιακά εργαζόμενε. Θα εγκρίνετε μέτρα για να βελτιώσετε τι ειδικές εργασία σε άλλου τομεί όπου υπάρχει μεγάλη επισφάλεια και κυρίω απασχολούνται οι γυναίκε, όπω για παράδειγμα οι καθαρίστρε στα ξενοδοχεία. Δύο λεπτά για την απάντησή σα. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι, φυσικά. Πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Και θα ασχοληθούμε. Ήδη έχω συζητήσει με τον υποψήφιο επίτροπο Σμιτ για την πραγματικότητα για τα θέματα αυτά. Αναφέρθηκα και πάλι σε αυτή την ειδική ομάδα. Εκεί μπορούμε να εργαστούμε μαζί με άλλους, με διάφορους συναδέλφους επιτρόπους, με διάφορους αλμοδιώτες, δηλαδή οι οικιακά εργαζόμενες, ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας τους και για τη σύμβαση του Διεθνούς ε, Γραφείου Εργασίας. Όλα αυτά είναι στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Απασχόλησης. Αλλά θα υπάρχει κάποιος ε, σύνδεσμος στις υπηρεσίες αυτού του Επιτρόπου που θα ασχολείται με τις εργαζόμενες αυτές. Ναι. Τα προβλήματα που αναφέρατε, οπωσδήποτε, θα με απασχολήσουν. Συλλογματική ερώτηση, παρακαλώ ένα λεπτό. Ξέρουμε ότι πολλές από τις οικιακά εργαζόμενες είναι μετανάστριες. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης και αυτό είναι σχεδόν αόρατο. Είναι σχεδόν αόρατες αυτές οι γυναίκες. Θα λάβετε μέτρα ούτως ώστε το γεγονό ότι είναι μετανάστριες να μην τις κάνει πιο ευάλωτες και να μην υποστούν ε, περαιτέρω βλάβη τα ήδη περιορισμένα δικαιώματά τους όσον αφορά τη συνταξιοδότηση. Τώρα που περνάει σε ιδιωτικούς φορείς η συνταξιοδότηση ή που γίνεται η που γινεται ακόμη και της κοινωνικής προστασίας. Ε, τι πιστεύετε για ένα ευρωπαϊκό σύστημα συντάξεων για όλους, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ήδη ψαλίδα μεταξύ ανδρών και γυναικών στους μισθούς και τις συντάξεις. Απάντηση. Όπως ξέρετε υπάρχει η οδηγία για την ισότητα που προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διακρίσεων σε όλους τους τομείς της ζωής και ένας από τους τομείς όπου υπάρχουν προβλήματα είναι οι συνθήκες πρόσβασης στην απασχόληση και οι συνθήκες εργασίας. Πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Αυτό θα είναι ο στόχος μου. Εντάξει, πιο εύκολο να το πεις παρά να το κάνεις. Αλλά υπάρχουν ήδη τα μέτρα για την προστασία. Το θέμα είναι πώς θα ελέγξουμε ότι γίνεται σωστά η εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Και φυσικά θα συνεργαστώ και με άλλους συναδέλφους επιτρόπους και για αυτό το θέμα. Κυρία Φριτζόν. Ευχαριστώ. Στα ειδικά θα κάνω την ερώτησή μου, κυρία Ντάλη. την τελευταία δεκαετία έχουμε διαπιστώσει ε, στεναρή αντίσταση ε, στα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών. Και ένας δείκτης για την ισότητα των φύλων δείχνει ε, ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές και ανισότητες μεταξύ των φύλων ακόμα. Πρόσφατα υπήρξε και έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έδειχνε ότι οι εξελίξεις είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα για διάφορους ε, λόγους. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, υπάρχουν μόνο κούφια λόγια, έτσι μια ρητορική, σε άλλες περιπτώσεις μέτρα που εφαρμόζονται. Εσείς βλέπετε να έχουν οπισθοδρομήσει τα γυναικεία δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εγώ θέλω να πω στι κόρες μου ότι αυτά ε, θα πρέπει να τα καταπολεμήσουμε και θα το κάνουμε. Ποια θα είναι η πρώτη σας πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή. Απάντηση. Εργαζόμαστε για την ισότητα των φύλων. Και βλέπετε πόση σημασία αποδίδει σε αυτά τα θέματα η εκλεγμένη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να φροντίσουμε όχι απλώς να προστατεύονται, αλλά να ενισχύονται τα γυναικεία δικαιώματα. Βέβαια, όπως βλέπετε και από τον αριθμό των επιτρόπων, ε, ε, αναζητούμε μια ισορροπία μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έχουμε και επίτροπο που είναι επιφορτισμένη με αυτό το χαρτοφυλάκι. Ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι ύψιστη προτεραιότητα της εκλεγμένης Προεδρού Φόντερ Λάιεν και για το λόγο αυτό υπάρχει ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο και επίτροπος για τα θέματα ισότητας. Άρα ε, ε, ακριβώς θέλουμε να εστιάζει ένας επίτροπος, μία επίτροπος σε αυτά τα θέματα και στα προβλήματα τα οποία εσείς αναφέρατε. Και η στρατηγική για την ισότητα των φύλων ε, που επίκειται αντιμετωπίζει κάποιες από τις καταστάσεις που εσείς περιγράφετε. Ένα λεπτό για τη συμπληρωματική σας ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες οφείλουν να αυτοπροσδιορίζονται και να... Ε, ε, ε, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια πολιτική για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της δυσμενούς αντιμετώπισης στους χώρους εργασίας. Ποια είναι τα μέτρα αυτά που εσείς προτείνετε έτσι ώστε οι γυναίκες να είναι αυτάρκεις οικονομικά. Οικονομική ανεξαρτησία είναι πραγματικά ε, θεμελιώδους σημασίας. Κάθε γυναίκα θα πρέπει να είναι σε θέση, να είναι νομικά ανεξάρτητη, να συντηρεί τον εαυτό της και αυτή τη στιγμή μια γυναίκα είναι οικονομικά ανεξάρτητη, αλλάζουν και τα πράγματα και πραγματικότητες τις οποίες ζει. Για παράδειγμα, όταν είσαι οικονομικά ανεξάρτητη, ε, μπορείς να επιλέξεις να φύγεις από μια σχέση ε, στην οποία εφίστασε διακρίσεις και καταχρήσεις ή κακομεταχείριση, γιατί δεν εξαρτάσαι οικονομικά από το δράστη ε, Έτσι, έχουμε περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες στην αγορά εργασίας και θα πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη κατάρτιση και εκπαίδευση για τις γυναίκες Υπάρχει μεν αυτή η κατάσταση σήμερα, αλλά πολλέ ε, είναι οι γυναίκες που παραμένουν εξαρτημένες οικονομικά. Η κυρία Φίλιψ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Επίτροπε, ε, υποψήφια επίτροπε, είπατε πως είστε ικανοποιημένοι με την οδηγία περί ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής. Ωστόσο, δέκα μέρες μόνο προβλέπονται ώστε οι γονείς, οι πατέρες μάλλον, να φροντίσουν τα παιδιά τους και, αυτά δεν, και αυτές δεν είναι υποχρεωτικές. Και ακόμα και αν το επιλέξουν οι, οι γονείς ε, φοβούνται ότι μπορεί να πέσουν από την, ε, στη φτώχεια εάν χρησιμοποιήσουν αυτό το είδους την άδεια, διότι δεν είναι αμοιβόμενοι. Ε, θα πρέπει λοιπόν όλοι οι άνθρωποι αλλά και οι γονείς κάθε φίλου και η ΛΟΑΔΜΑ να μπορούν να πάρουν άδεια για να φροντίσουν τα παιδιά τους. Τι θα κάνετε ώστε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα της ισορροπίας, τι θα προτείνετε στις οικογένειες, ώστε μάλλον οι οικογένειες να μην αντιμετωπίζουν την φτώχεια όταν ζητούν άδεια. Τι θα κάνετε ώστε τα κράτη-μέλη να προσφέρουν αμοιβή, αξιοπρεπή αμοιβή για αυτό του είδος την άδεια. Δύο λεπτά για την απάντησή σας. Ναι, ε, είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινήσατε με με αυτή την οδηγία που είπα ότι πάει προς τη σωστή κατεύθυνση και γι' αυτό είπα ότι θα παρακολουθώ τα κράτη-μέλη ώστε να δούμε πώς την εφαρμόζουν. Και Ίσως και να κάνουμε και σεμινάρια και παρουσιάσεις έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι ότι πρόκειται για προστιθέμενη αξία για το, για το χώρο εργασίας όταν ισχύουν τέτοιου είδους μέτρα. Βεβαίως θέλουμε να κάνουμε περισσότερα και όπως ανέφερα σε τρία χρόνια θα αναθεωρηθεί αυτή η οδηγία. Και πιστεύω πως ε, οι εργοδότες θα έχουν κατανοήσει πια πως πρόκειται για κάτι το θετικό. Πάντως, οποτεδήποτε κάνεις κάτι το οποίο σχετίζεται με τις εργασιακές σχέσεις, θέλεις οι εταίροι σου να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν την αξία. Και αυτό είναι κομμάτι του κοινωνικού διαλόγου. Όσο περισσότερο λοιπόν βοηθήσουμε τους κοινωνικούς εταίρους να κατανοήσουν την προστιθέμενη αξία που έχουν οι καλές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους, ότι δηλαδή εργαζόμενοι μέσα σε καλές, καλύτερες συνθήκες εργάζονται καλύτερα, είναι πιο ήρεμοι, αποδίδουν περισσότερο, δηλαδή είναι προς όφελος των, εργοδοτών να ισχύουν πολύ καλές εργασιακές συνθήκες, τόσο το καλύτερο. Όλα όσα είπατε λοιπόν είναι αληθή και θα θα συζητήσω όλα αυτά και με τον υποψήφιο Σμιτ όταν θα μιλάμε για τις συνθήκες απασχόλησης. Αλλά βεβαίως υπάρχει και η προοπτική της ισότητας εδώ. Να, διακόπτη πρόεδρος. Επερώτηση. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Η παραδοσιακή ε, μοιρασιά εργασίας ε, με τις ε, γονικές ευθύνες αλλάζει, αλλά πολύ αργά. Έχουμε μιλήσει για αυτά τα πράγματα, αλλά για πολύ χρόνο μιλήσατε για σεμινάρια και συζήτηση με τους συναδέλφους τους επιτρόπους. Η νομοθεσία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Τι θα κάνετε συγκεκριμένα ώστε να ξεπεραστεί αυτή η αδικία που θα είναι περισσότερο από ότι απλά και άλλα λόγια και σεμινάρια. Χωρίς μικρόφωνο. Μάλιστα. Πρέπει να επαναλάβω ότι μόλις θα αναθεωρήσουμε και θα εξετάσουμε, αξιολογήσουμε μάλλον το πώς λειτουργήσε η οδηγία και εάν υπάρχει πεδίο, μάλλον θα υπάρχει πεδίο για να την ε, αναθεωρήσουμε, τότε θα εξετάσουμε τις προτάσεις που υποβάλλετε εσείς. Ευχαριστώ. Η κυρία Σεμέδο, την ερώτησή σας για ένα λεπτό. Λοιπόν, θα μιλήσω γερμανικά. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, κυρία Ντάλη, η ερώτησή μου έχει να κάνει με την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Θα ήθελα να πω περισσότερα για αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε τι συγκεκριμένε δυνατότητε. θεωρείτε ότι υπάρχει στη Σύμβαση τη Ένωση, ώστε να αντιμετωπιστεί η βία κατά των γυναικών να θεωρηθεί ενωσιακό έγκλημα. Πρέπει επίση να βοηθήσουμε τα θύματα να μπορέσουν να επανέλθουν στην κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γυναίκε δηλαδή οι οποίοι ήσαν θύματα βίας ε, ε, αλλά και γυναίκες για παράδειγμα που έχουν πάθει καρκίνο και έχουν επιβιώσει. Αλλά μετά έχουν χέρες, για παράδειγμα για να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά για την απάντησή σας. Η βία κατά των γυναικών να θεωρηθεί ενωσιακό έγκλημα Χρειάζεται ομοφωνία για να γίνει. Το λένε και οι κατευθυντήρες γραμμές. Αλλά πρώτα θα εστίαζα περισσότερο στην επικύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Νομίζω ότι αυτός θα είναι ο χρυσός κανόνας, αυτή θα είναι η βασική προδιαγραφή. Ας ε, εστιάσουμε λοιπόν σε αυτό. Αλλά να γίνει ενωσιακό έγκλημα, όπως είπα, η βία κάτω των γυναικών, ε, όπως είπα, χρειάζεται ομοφωνία. Βεβαίως μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο τις γυναίκες μέσω ενίσχυσης οδηγίες για τα δικαιώματα των θυμάτων. Εκεί θα συνεργαστώ με τον υποψήφιο επίτροπο Ρεντέρθ. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα νομοθετικά για να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών. Αλλά για μένα το πιο βασικό τώρα είναι η επικύρωση από την Ένωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Συμπληρωματική ερώτηση ένα λεπτό. Θα κάνετε και μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης ε, για την ενδογενειακή βία με επαρκείς πόρους. Ευαισθητοποίηση και για τους νέους και τους πιο ηλικιωμένους να έχουν υπόψη τους και τα θύματα δηλαδή, ποια είναι τα δικαιώματά τους. Γιατί Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει κανείς να μην καταπιέζεται και κανείς να μην είναι θύμα βίας. Απάντησε. Ναι, φυσικά. Ναι, θα συμπεριληφθεί. Στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων και θα συμπεριλάβουμε και την βία στο ίντερνετ κατά των γυναικών. Τα σημεία που αναφέρατε. Θα τα συμπεριλάβουμε. Γιατί η στρατηγική αυτή με πολύ αποφασιστικό τρόπο αντιμετωπίζει τα θέματα βίας κατά των γυναικών και επίκειται η έκδοσή της. Τελευταία ε, ομιλήτρια, κυρία Γιαρόκα, με τη δική σας ερώτηση ολοκληρώνεται γύρω στον Ένα Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, συγχαρητήρια. Και μετά ε, από την Οδύνη ε, της καταπληκτικής γυναίκας από τη Μάλτα, της Δάφνε ε, Καρουάνα Γαλίτσια. Χαίρομαι που βλέπω άλλη μια θαραλέα γυναίκα από τη Μάλτα. Μιλήσατε για το συνταξιοδοτικό και το μισολογικό χάσμα. 16% στους μισθούς η ψαλίδα και 36% στις συντάξεις. Ε, θα κάνετε κάποια συγκεκριμένα βήματα από αυτόν. Δύο λεπτά για την απάντηση. Προφανώς. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να βρούμε στις πρώτες 100 ημέρες ένα τρόπο μέτρησης. Θα καταθέσω ε, αυτό το μέτρο για τη διαφάνεια ε, στις αμοιβέ. Από εκεί και πέρα μπορούμε να ε, μετρήσουμε ποια είναι αυτή η ψαλίδα στους μισθούς και τις συντάξεις ακριβώς. Είναι από τα πρώτα πράγματα που πρόκειται να κάνω και από τους πρώτους τομείς που έχω εντολή να ασχοληθώ και να εργαστώ. Αυτό δείχνει πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα και πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ε, εξετάζει με πολύ μεγάλη προσοχή, του δίνει πολύ μεγάλη σημασία και φυσικά θέλουμε να έχουμε και αποτελέσματα. Γιατί είναι απαράδεκτο να υπάρχει τέτοια διαφορά. 36% συντάξει. Αυτά είναι κατάλοιπα όλων αυτών που είπαμε σήμερα. Για το πόσο έχει ο εργασιακός βίος μιας γυναίκας και ο κύκλος αυτός. Η πρόοδος της σταδιοδρομία της πολλές φορές διακόπτεται. Γιατί εργαζόμαστε για λιγότερες ώρες, έχουμε μειωμένο ωράριο λόγω των οικογενειακών αναγκών ή καμιά φορά όταν μια γυναίκα είναι σε άδεια μητρότητας ή εργάζεται ε, σε μειωμένο ωράριο, χάνει ε, μια προαγωγή και χάνει και την ανέλυξή της. Δηλαδή, υφιστάμεθα αυτή τη τιμωρία, επειδή είμαστε γυναίκες, έχουμε παιδιά, θέλουμε να κάνουμε παιδιά και θέλουμε και να εργαστούμε. Είναι σημαντικό να συνεισφέρουμε με τη δουλειά μας. Αλλά μετά ερχόμαστε αντιμέτωπες με αυτές τις πραγματικότητες και αυτές τις διαφορές. Ε, συμπληρωματική ερώτηση για ένα λεπτό παρακαλώ. Αυτές οι διαφορές πραγματικά ε, ρίχνουν ε, περισσότερο στη φτώχεια ε, τις γυναίκες και τα παιδιά. Και θέλω να σας ρωτήσω <laughs> για τις γυναίκες και για τους φτωχούς. 120 ε, εκατομμύρια είναι οι ε, φτωχοί. η Ρωμά είναι μόνο 16 εκατομμύρια. Αλλά για όλους αυτούς που δεν έχουν δουλειά ε, είναι όνειρο το χάσμα το μισθολογικό. Και τα γκέτο δεν είναι μόνο στην Ανατολική Ευρώπη. Θα τα συμπεριλάβετε όλα αυτά στην πολιτική σας. 30.000, 80.000 άνθρωποι σε διάφορους οικισμούς και ε, χρειάζεται αντιμετώπιση. Υπάρχουν χάρτες του 2016 που τα δείχνουν όλα αυτά. Μία από τις πρώτες μου επισκέψεις θα είναι σε καταβλισμό Ρωμά. Οι Ρωμά υφίστανται τις περισσότερες διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 61%. Όπως γνωρίζετε υπάρχει μια στρατηγική πλαίσιο για τους Ρωμά με τέσσερις προτεραιότητες, εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία και στέγη. Ξέρετε ότι λύγει προσεχώς αυτό το πλαίσιο αυτή τη στρατηγική επίσης θα την ε, αξιολογήσουμε, θα την αναθεωρήσουμε. Ε, Θέλω να επισκεφτώ ένα τέτοιο καναβλισμό για να καταλάβω καλύτερα και να γνωρίζω περισσότερο τι αξιολογώ και τι αναθεωρώ και πώς θα προχωρήσουμε καλύτερα και τι συνέχεια θα δώσουμε. Και το επόμενο πλαίσιο μετά το 2020 θα εστιαστεί περισσότερο στις διακρίσεις εις βάρος των Ρωμά, στον αντιτσιγκανισμό σας διαβεβαιώ ότι θα γίνει πολλή δουλειά σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η τελευταία σας απάντηση. Κυρία Επίτροπε, <laughs> όμως δεν πρόκειται να βρείτε ησυχία γιατί θα σας ξαναδώσουμε το λόγο για πέντε λεπτά για την τελική σας ε, τοποθέτηση, τα καταληκτικά σας σχόλια. Παρακαλώ. So thank you for the exchange and for... Ευχαριστώ για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων για τις σημαντικές ερωτήσεις που μου θέσατε. Και αυτό που φαίνεται από αυτά που συζητήσαμε είναι ότι η ισότητα ποτέ δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Ξέρω ότι με εμπιστεύεστε. Μάλλον καλύτερα. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Δεν ήθελα να πω αυτό. Ξέρω ότι αν με εμπιστευτείτε για να αναλάβω το ρόλο επιτρόπου θα πρέπει να αντιμετωπίσω πολλές δύσκολες προκλήσεις για να, για να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Και προσβλέπω στις περαιτέρω συζητήσεις για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Καταλήγοντας, να σας πω κάτι προσωπικό. Όποτε πήγα σε δημοτικό, σε νηπιαγωγείο ή σε βρεφονιπιακό σταθμό ως υπουργό, πάντα έβλεπα πως τα μικρά παιδιά έρχονται σε επαφή και παίζουν μεταξύ τους χωρίς να κάνουν διακρίσεις. Δεν καταλαβαίνουν καν τι σημαίνει διάκριση, δεν αποκλείουν κανένα. Τα παιδιά παίζουν με τα άλλα παιδιά παρά το πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι. Δεν κάνουν διακρίσεις. Δεν μισούν. Τα παιδιά μας ε, διδάσκουν τι σημαίνει αγάπη ανεφόρων. Οι διακρίσεις είναι κάτι που τους περνάει αργότερα στη ζωή. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε ούτω ώστε η κοινωνία να ξεπεράσει τα στερεότυπα, να ξεπεράσει τις διακρίσεις που πολλές φορές οφείλονται στα προσωπικά χαρακτηριστικά. Είμαστε πιο ισχυροί αν είμαστε μια ένωση κρατών μελών. Είμαστε πιο ισχυροί ως κοινωνίες με τόσες διαφορές όταν όλα μας τα μέλη δεν εξαιρούνται από τίποτα και όταν ε, όλοι έχουν την ίδια αξία για όλους. Θέλω να βοηθήσω όλες τις φιλετικές μειονότητες, εθνικές μειονότητες, με ιδιαίτερη προσοχή στους Ρωμά. Επίσης ε, και όλες τις θρησκευτικέ και μη θρησκευτικέ ε, κοινότητες. Όλα τα άτομα που υφίστανται διακρίσεις για λόγους ε, της ηλικίας τους, για λόγους αναπηριών ή για λόγους εξωτερικού προσανατολισμού. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε αρκετή ισότητα για όλους. Πρέπει να γίνει πραγματικότητα που να την βιώνουν όλοι στην καθημερινότητά τους. Όπως είπε ο Νέλσον Μαντέλα, που θα συνεχίσει να είναι πάντα ο δικός μου, κανείς δεν γεννιέται με μίσος για τους άλλους, λόγω του χρώματος, του δέρματός του, ή της προέλευσής του, ή της θρησκείας του. Τα άτομα μαθαίνουν να μισούν. Αλλά ε, εφόσον μαθαίνουν να μισούν μπορούν επίσης να διδαχθούν να αγαπούν. Γιατί η αγάπη είναι πιο φυσιολογικό συνέστημα για την ανθρώπινη ψυχή από το αντίθετό της. Σας ευχαριστώ πολύ. So, uh, Λοιπόν, Αγαπητή υποψήφοι επίτροπε, κυρία Ντάλη, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα καταφέραμε. Όπως βλέπετε, ήταν πολύ σκληρή δουλειά όλες αυτές οι ερωτήσεις και το μεγάλο, το μακρύ το ταξίδι της ισότητας. Και βλέπουμε ότι η ισότητα είναι ένα θέμα που χρειάζεται μια επίτροπο ε, σκληρή, στεναρή, έτοιμη, αποφασισμένη, που δεν είναι ε, μόνο έτοιμη να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο, αλλά που να καταλαβαίνει επίσης τι σημαίνει να εφίστασε διακρίσεις και να υποφέρεις από τις ανισότητες. Και ακούσαμε τόσους πολλούς από τόσες πολιτικές ομάδες, ένα ευρύτατο φάσμα ερωτήσεων που καλύπτουν όλες τις πολιτικές ομάδες. Και πάνω απ' όλα και μιλώ εξ ονόμα της Επιτροπής ΦΑΜ, Δικαιωμάτων των Γυναικών, οι γυναίκες που υφίστανται ανισότητες στην καθημερινή τους ζωή, άκουσαν απαντήσεις ε, σαφείς και ρεαλιστικές για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Τι θα κάνουμε στο μέλλον. Από τη Μελλοντική Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχοληθήκατε με τα θέματα του μισθολογικού χάσματος που είναι όνειδος γιατί δεκαετίες ολόκληρες βλέπουμε ότι αργούμαστε, ε, κινούμαστε συγγνώμη, με τόσο αργούς ρυθμούς και θέλουμε διαφάνεια για να εφαρμόσουμε μέτρα έτσι ώστε οι γυναίκες να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους άνδρες. Αναφερθήκαμε στο θέμα της βίας κατά των γυναικών, τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που θα πρέπει πραγματικά να είναι ζωντανή και πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση ακούσαμε σε τόσες πολλές χώρες και τι δικαιολογίε ακούμε από κυβερνήσεις, από τον οποιοδήποτε για να μην κάνουν αυτά που οφείλουν να κάνουν. Επίσης αναφερθήκατε ε, στη στρατηγική για το φύλλο που χρειαζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα μέτρα, γιατί Ωραίο είναι να βάζεις ένα λιθαράκι, μία ψηφίδα σε ένα του... αλλά θα πρέπει όλη η εικόνα να αποκτήσει η ζωή. Και επίσης ασχοληθήκαμε και με ένα πλήθος άλλων θεμάτων που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ισότητα ανδρών και γυναικών και ασχοληθήκαμε και με τις διακρίσεις που τις βλέπουμε σε κάθε τομέα της ζωής. Με τούτα εδώ τα λόγια θα ήθελα απλώς να σας συγχαρώ για αυτό το μαραθώνιο ερωταπαντήσεων ε, που κάλυψαν όλα αυτά τα θέματα. Και τώρα ήρθε η ώρα των συντονιστών να αποφασίσουν. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σας ευχαριστώ και πάλι για το μαραθώνιο αυτό και την επίδοσή σας και θα δώσω μες το λόγο στην συνπρόεδρό μου, την κυρία Νικόλ Σόνοβα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ντάλη. Θα πρέπει να πω ότι ήσασταν πολύ, πολύ πειθαρχημένοι, πολύ καλοί στο χρόνο σας. Αυτό τα καταφέρατε πολύ καλά. Εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης θα πρέπει να σας πω ότι το δικό σας χαρτοφυλάκι είναι τόσο ευρύ και τα σχέδιά σας τόσο φιλόδοξα που θα θέλαμε πραγματικά να συνεργαστούμε μαζί σας για όλα σας αυτά τα φιλόδοξα ε, σχέδια. Όμως πιστεύω πως ε, πρέπει να υποσχόμαστε μόνο αυτά που μπορούμε πραγματικά να καταφέρουμε γιατί ο κόσμος περιμένει, έχει τεράστιες προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Βρυξέλλες. Και όσον αφορά νέες πρωτοβουλίες νομίζω πως θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσουμε πώς θα καταφέραμε με την εφαρμογή των παλιών πρωτοβουλειών ώστε, ε, γιατί έτσι για να είμαστε ειλικρινείς δεν τα έχουμε καταφέρει παντού ε, υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουμε ε, τους αναπήρους που υποφέρουν από διακρίσεις φρικτές. Δεν μπορούν να βγουν στο δρόμο, δεν μπορούν να πάνε στο σινεμά, στο θέατρο, ε, δεν μπορούν να βρουν δουλειά, ε, δεν μπορούν να τα καταφέρουν στην αγορά εργασίας. Οι εταιρείε προτιμούν να ε, πληρώνουν ε, πρόστιμα παρά να απασχολήσουν κόσμο με αναπηρίες. Επίσης πρέπει να μιλάμε και για τους ανθρώπους ανά των 50 στην αγορά εργασίας που αντιμετωπίζουν τεράστιες διακρίσεις στα διάφορα κρατημέλη και αυτή είναι μια, ε, μια γενεά σάντουιτς που πρέπει να την αναφέρουμε όταν μιλάμε για ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για νέους ανθρώπους και με μικρά παιδιά. Πρέπει να μιλάμε και για τους ανθρώπους άνω των 50 που ε, είναι από την άλλη πλευρά και ε, αρχίζουν να γίνονται ε, ηλικιο... περισσότερο ηλικιωμένοι. Επίσης έχουμε κοινωνικό αποκλεισμό σε πολλά κράτη-μέλη, έχουμε τις κοινότητες Ρωμά όπου σε πολλά κράτη-μέλη ανοιχτά γίνονται διακρίσεις κατά αυτών των κοινοτήτων, πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία και δεν καταφέρουν να τελειώσουν ούτε καν το δημοτικό δημοτικό σχολείο ε, δεν μπορούν, και ενώ φτάνουν στα 16 μπαίνουν στα ειδικά σχολεία και δεν μπορούν ούτε να γράψουν ούτε να διαβάσουν και θέλουμε εμείς να τους βάλουμε στην αγορά εργασίας. Είμαι, χαίρομαι που η κυρία Νταλή θα έρθετε και σε μια αντιπροσωπεία της επιτροπής μας που θα πάει στη Σλοβακία και θα επισκεφθεί τις κοινότητες της Ρωμά να πάψουν πια οι διακρίσεις κατά τον Ρωμά. Ευχαριστώ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται η ακρόαση αυτή. Χαίρετε.